Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φιλοξενούμενοι. Τις εξοχότητές σας, τους πρεσβευτές, επίσης σας καλωσορίζω στην Επιτροπή μας. Θερμό καλωσόρισμα λοιπόν. Και τον κύριο Όλιβερ Βερχέη καλωσορίζω, υποψήφιο για θέση Επιτρόπου για θέματα γειτονίας και διεύρυνσης. Κύριε Βερχέη, καλώς ήρθατε στην Επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων. Χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ σήμερα διότι αυτή είναι πολύτιμη ευκαιρία για μας για διάλογο και πρώτο σημαντικό βήμα για επικοδομητική καρποφόρα συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι σίγουρος ότι θέλετε να έχετε στενές διασυνδέσεις και διάδραση με μας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο μέλλον. Συνάδελφοι, να υπενθυμίσω κάτι. Σκοπός ακροάσεω είναι το Κοινοβούλιο να αξιολογήσει τον υποψήφιο επίτροπο και αυτό βάσει των γενικών του ικανοτήτων, γνώσεων, το κατά πόσο ασθενίζεται το ευρωπαϊκό εγχείρημα και κατά πόσο προσωπικά ανεξάρτητο. Θα αξιολογήσουμε τη γνώση, τις γνώσεις για το χαρτοφυλάκιό του και τι δυνατότητε που έχει να επικοινωνεί. Στι 13 Νοεμβρίου λάβαμε την απαντήση του κ. Βερχέη στις γραπτές μα ερωτήσεις διανεμήθησαν σε όλα τα μέλη, σε όλες τις γλώσσες και έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. Επιτρέψτε μου τώρα, εν συντομία, να σας αναφέρω πώς θα διεξαχθεί η ακρόαση, που βεβαίως διοργανώθηκε σύμφωνα με το εσωτερικό κανονισμό του Κοινοβουλίου για να εξασφαλίσουμε δίκαιε και ισότιμε συνθήκε για όλου του υποψήφιου επιτρόπου να παρουσιαστούν και να παρουσιάσουν τι απόψει του. Καταρχά, ο υποψήφιο επίτροπο θα κληθεί να προβήσει μια ανακτήρια ομιλία που δεν θα κρατήσει πάνω από 15 λεπτά. Μετά από αυτή την εισαγωγή θα υπάρχει χρόνος για 25 ερωτήσεις από πλευράς μελών. Στον πρώτο γύρο θα έχουμε τις ερωτήσεις που βληθούν από τους ε, αρχηγούς των πολιτικών ομάδων και στο δεύτερο γύρο θα μιλήσουν 18 μέλη σύμφωνα με τις ποσοστώσεις που έχουν δοθεί σε διάφορες πολιτικές ομάδες και θα ακούσουμε και εκπροσώπους των μη εγγεγραμμένων μελών. Αυτά τα, αυτές οι πεντάλεπτες χρονοθυρίδες ερωταπαντήσεων απαντήσουν στο εξή. Κάθε μέλος έχει ένα λεπτό χρόνο στη διάθεσή του να υποβάλει την ερώτησή του, ερώτησή της. Μετά θα ακολουθήσει η δίλεπτη απάντηση από τον υποψήφιο επίτροπο. Μετά, αν χρειαστεί, υπάρχει δυνατότητα το ίδιο μέλος αμέσως να υποβάλει σημαντική ερώτηση, το πολύ για ένα λεπτό. Και τέλος, ο υποψήφιος επίτροπος μπορεί εκ νέου να δώσει απάντηση ενός λεπτού στην εν λόγω ε, συμπληρωματική ερώτηση να υπενθυμίσω στους ότι η συμπληρωματική ερώτηση μας σχετίζεται στην απάντηση υποψηφίου επιτρόπου στην πρώτη ερώτηση που χρησιμοποιηθεί σαν ευκαιρία για θήξη ε, θυγούν άλλα θέματα. Μετά ο υποψήφιος επίτροπος θα έχει πέντε λεπτά για να ολοκληρώσει, τη, να κάνει δευτερεύουσα παρέμβασή του. Έχουμε τρει ώρε στη διάθεσή μα. Παρακαλώ όλοι για να προλάβουμε να μιλήσετε στο χρονικό διάστημα σας διαθέσουμε. Αν μιλήσετε παραπάνω από το χρόνο σας, οι συνάδελφοι θα αφαιρέσουν χρόνο ομιλίας από άλλο συνάδελφό τους. Η διερμηνία εξασφαλίζεται προς 23 γλώσσες. Αυτή η ακρόαση μεταδίδεται ζωντανά από την ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου στη διαδίκτυο και είναι δυνατότητα να, να έχει κανείς βίντεο σκόπηση της ακρόασης στην ίδια ιστοσελίδα. Αυτά από την πλευρά μου εν είδη εισαγωγή. Αγαπητέ υποψήφιο επίτροπε, αγαπητέ κύριε Βερχέ, έχετε τώρα το, το λόγο για την ενακτήρια δήλωσή σα που μπορεί να κρατήσει μέχρι 15 λεπτά και έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Τιμή για μένα που έχω τη δυνατότητα ως υποψήφιος ε, επίτροπος για θέματα γειτονίας και διεύθυνση να σας παρουσιάσω σήμερα το όραμά μου για τις μελλοντικέ μας σχέσεις με τους γείτονες και τους εταίρους. Ε, καταρχάς, επιτρέψτε να πω μερικά λόγια για τον εαυτό μου, που ίσως σας βοηθήσουν να καταλάβετε ποιο είναι το όραμά μου για το έργο που έχω μπροστά μου, αν τελικά επικυρωθεί ο διορισμός μου. Γεννήθηκα στην κομμουνιστική Ουγγαρία, τα μέλη της οικογένειας μου ήταν θύματα δίωξης μετά το 1956, η επανάσταση που συνεθλίβε από το Σοβιετικό στρατό και ακολούθησε το καθεστώς και από τότε μορφώθηκε η συνείδησή μου από αυτά τα γεγονότα από πολύ νωρίς. Η πτώση του κομμουνισμού άνοιξε το δρόμο για τις χώρε κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης να ξανενωθούν με την ελεύθερη Ευρώπη. Εγώ ανήκω στη νέα γενιά των Ούγγρων, ε, οι οποίοι υλοποίησαν αυτό το όνειρο. Η διεύρυνση του 2004 ήταν ένα όνειρο που αληθεύτηκε για μας. Έκτοτε πάντα εργαζόμουν για να είναι μια επιτυχία αυτή. Υπηρέτησα τη χώρα μου και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορες ε, θέσεις. Ε, έμαθα ότι τα συμφέροντα των κρατών μελών και της ενώσεως ίσως να αποκλίνουν για κάποια ζητήματα, αλλά απότερος σκοπός είναι κοινό να οικοδομήσουμε ισχυρή και επιτυχή Ευρώπη προς όφελος όλων. Κατευθυντήρια αρχή που πάντα ακολουθούσα ήταν η σύνθεση Στόχος μου είναι να βρω κοινό τόπο και σχέσεις μεταξύ των διαφόρων θέσεων και να δημιουργώ λύσεις οι οποίες ε, λειτουργούν για όλους, παραδείγματο χάρη, όταν υπηρέτησα σαν ε, διοικητικό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήμουν υπεύθυνο που δημιούργησα το... την πατέντα της Ευρωπαϊκής Ενώσεω, το δίπλωμα βεστιτεχνία. Η Ουγγαρία ήταν κατά αυτού αρχικά, όμως κατάφερα να τονίσω ποια είναι τα ωφέλη που υπάρχουν και σε πολλού άλλου και δημιουργήσαμε την ευρωπαϊκή, το ευρωπαϊκό αυτό, ε, αυτή την πατέντα που ήταν επιτυχές ε, αποτέλεσμα. Δεν θέλουμε να επιλέξουμε μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών συμφερόντων για να οικοδομήσουμε την Ευρώπη. Θέλουμε να βρούμε τις λύσεις που συνθέτουν και συγκεράζουν τις διάφορες θέσεις. Θέλω να συνεχίσω βάσει αυτής της αρχής Σαν Ευρωπαίος Επίτροπος, αν επικυρωθεί η θέση μου, θα αποτελέσω γέφυρα μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκπροσωπεί τους πολίτες άμεσα, ε, να ενώσω με το Συμβούλιο που εκπροσωπεί τα κράτη-μέλη και να ενώσω και τις θέσεις αυτές με τις θέσεις των γειτονικών χωρών. Η γειτονιά μας είναι πολύ σημαντική, στατική σημασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μοίρα μας συνδέεται και επηρεάζεται σημαντικά από τη μοίρα των γειτόνων μας Υπάρχει μεγάλη διαφορά εξέλιξης και ανάπτυξης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και γειτόνων. Στόχος μου θα είναι να μειώσω αυτό το κενό εκμεταλλευόμενος τις κρυφές δυνατότητες που έχουν οι περιοχές. Κατά τη διάρκεια τη ε, θητεία μου θέλω να ενισχύσω το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω για την πρόθεση τη ασφάλεια, τη σταθερότητα και για την πρόθεση τη ε, ευημερία σε μια γειτονιά που αλλάζει και δημιουργεί προκλήσεις. Θέλω να υποστηρίξω τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη που θα στηρίζεται σε μια λειτουργούσα οικονομία της αγοράς με ισχυρούς δημοκρατικούς θεσμούς, να επικρατεί το κάτω δικαίου και θεμελιώδεις ελευθερίες. Ε, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα μείνει εκτός και πίσω Γι' αυτό θέλω να βοηθήσω τους εταίρους μας να ενισχύσουν την κοινωνική διάσταση της οικονομίας τους συγχρονισμένοι με την οικονομική τους ε, ανάπτυξη. Εάν δεν επομιστούμε τις ε, ευθύνες μας, άλλοι θα πάρουν τη θέση μας. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ποιες είναι οι διαφορές πραγματικότητες και περιστάσεις που αντιμετωπίζουν οι εταίροι μας στη γειτονιά μας και πρέπει να του υποστηρίξουμε με, κατανά... με τις διάφορες συνθήκες που απαιτεί ο καθένας τα Δυτικά Βαλκάνια, η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία έχουν προοπτικέ αφή για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να βοηθήσουμε να ενστερνιστούν τι ευκαιρίε που παρουσιάζει αυτή η προοπτική, κάτι που στα μάτια μα είναι προ όφελό μα στρατηγικό. Άλλοι στρατηγικοί εταίροι, όπω είναι η Τουρκία, απομακρύνονται σαφώ από τι ευρωπαϊκέ αξίε και τι προδιαγραφέ. Θα πρέπει να δούμε πώ θα αντιμετωπίσουμε ε, αυτό το γεγονός πιο αποτελεσματικά. Κάποιοι εταίροι μας έχουν σημειώσει πρόοδο και έχουν κάνει μεταρρυθμίσεις άλλες ε, πλήττονται από, από κρίσεις όπως είναι στη Συρία στο Λίβανο, η Γεωργία, η Ουκρανία και η Μολδαβία προς Ανατολάς και στο Νότο, το Μαρόκο και την Ισία δείχνουν αποφασιστικότητα καμιά φορά υπό πολύ δύσκολες περιστάσεις να αντιμετωπίσουν το θέμα των μεταρρυθμίσεων. Άλλες χώρες δεν έχουν τόσο μεγάλη προθυμία και γι' αυτό ευφυής διαφοροποιημένη προσέγγιση σε όλο το χαρτοφυλάκιο είναι σημαντικό ούτω ώστε να μπορούμε να ξαγάγουμε σταθερότητα. Αξιότιμα μέλη, επιτρέψτε μου να προβούσε κάποια συγκεκριμένα σχόλια για κάθε περιοχή, ξεκινώντας από τα Δυτικά Βαλκάνια. Αυτή η περιοχή είναι αναπόσπαστο τμήμα της Ευρώπης και οι προοπτικές ένταξής της θα πρέπει να είναι κάτι αξιόπιστο. Αυτό είναι προς δικό μας γεωπολιτικό συμφέρον. Όμως πρέπει να στηρίξουμε και να επιταχύνουμε την προοδό αποτελεσματικότερα μέσω μιας διαδικασίας βάση επιδόσεων για κάθε χώρα θα πρέπει να εστιαστούμε επί του πραγματικού αντιχτύπου των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων, των επιτοπίων. Ε, θα πρέπει να προσμετρούμε την πρόοδο όσον αφορά την αύξηση της ευημερία και την ποιότητα διαβίωσης και την ελευθερία των ανθρώπων στην περιοχή. Αυτό είναι ο απότερος σκοπός της ενταξιακής διαδικασίας. Προτίθεμαι να αυξήσω το ρυθμό διαθροτικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων, εστιαζόμενο επί των θεμελιωδών στοιχείων, δηλαδή κράτος δικαίου, οικονομική ανάπτυξη, λειτουργία δημοκρατικών θεσμών και μεταρρύθμιση στον τομέα τη δημόσια διοίκηση. Έχω σε επαφή με όλα τα θεσμικά όργανα, τι επιχειρήσει και την κοινωνία των πολιτών για να πετύχω του εν λόγω στόχου. Θα συνεχίσω να υπερασπίζω με την πρόταση να ανοίξουμε ενταξιακέ διαπραγματεύσει με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Θα κάνω ό,τι μπορώ τους ώστε αυτό να συμβεί το συντομότερο δυνατό. Μεγάλοι Ευρωπαίοι ηγέτες επισκέφθηκαν τη Βόρεια Μακεδονία πριν το δημοψήφισμα για τη Συμφωνία των Πρεσπών και υποσχέθηκαν ότι αν πέρναγε οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις θα ξεκινούσαν. Η Αλβανία επίσης έχει εφαρμόσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο δικαστικό τομέα και στη δημόσια διοίκηση ανταποκρινόμενη στα αιτήματά μας. Με άλλα λόγια, αυτό που διακυβεύεται εδώ είναι η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή και πέραν αυτής. Θα εργαστώ επίση όταν να εντάξουμε καλύτερα την περιοχή στι βασικέ πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω ακόμα πριν την προσχώρησή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επί παραδείγματα, να εξασφαλίσουμε τα Δυτικά Βαλκάνια συνδέονται στενά με την συμφωνία μα, την πράσινη συμφωνία, την ψηφιακή μας, το ψηφιακό μα θεματολόγιο και όσον αφορά τα διευρωπαϊκά δίκτυα στι μεταφορέ και την ενέργεια θα υποστηρίξω όλες τις προσπάθειες προς καλέ γειτονικέ σχέσεις, την επίλυση των διμερών διαφορών θα συνεργαστώ με τον Ιωζεφ Μπορέλ, ούτω ώστε ο διάλογο μεταξύ, μεταξύ Βελιγραδίου και Πριστίνα να ολοκληρωθεί επιτυχώ το έτος 2020. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ετοιμαστεί για να, να δεχτεί τα μελλοντικά κράτη-μέλη. Από τη στιγμή θα πληρούνται οι συνθήκε. Όμω, ε, θεωρώ ότι μπορούμε και να συνδυάσουμε ε, και την εμβάθυνση με τη διεύρυνση. Αυτό έχει συμβεί συχνά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα συνεργαστώ με τον κύριο Μπορέλ για τις σχέσεις μας στο μέλλον με την Τουρκία που είναι βασικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πάρα πολλούς ε, τομείς. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε τις σχέσεις μας για να υπηρετούμε καλύτερα τα συμφέροντά μας. Η Τουρκία εξακολουθεί να διαδραματίζει κομβικό ρόλο, εξακολουθεί να φιλοξενεί περίπου 4 εκατομμύρια πρόσφυγες, άρα δηλαδή θα πρέπει να να στηρίζουμε την Τουρκία σε αυτό το θέμα. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε βέβαια να κάνουμε τα στραβά μάτια σε αυτές τις πρόσφατες ανησυχητικές εξελίξεις. Πρέπει κυρίως να δούμε τις αρνητικές εξελίξεις στο κράτος δικαίου, στα ανθρώπινα δικαιώματα, η ε, Τουρκία έχει όλο και πιο προκλητική ε, εξωτερική πολιτική, προβαίνει σε παράνομες γεωτρήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Είχαμε και την παράνομη εισβολή στην ε, Συρία. Έτσι λοιπόν ε, θεωρούμε ότι δεν εστιάζεται η προσοχή ακριβώς στο να αντιμετωπιστεί η τρομοκρατία, ο Η επόμενη επιτροπή θα πρέπει να αρχίσει από κοινού με το Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο να εξετάζει το πώς μπορεί να σφυριλατήσει στρατηγική συνεργασία με βάση κοινέ αρχές και το υπάρχον πλαίσιο. Η ανατολική γειτονία. Στην ανατολική γειτονιά μας θέλω οι σχέσεις να ενισχυθούν ε, λαμβάνοντας υπόψη και τις διαβουλεύσεις που τρέχουν. Εγώ λοιπόν θα δουλέψω πάνω σε προτάσεις για, την, ε, για τους μακροπρόθεσμους στόχους της ανατολικής πολιτικής. Αυτά θα παρουσιαστούν από την Επιτροπή έγκαιρα πριν από την επόμενη συνάντηση για την εταιρική σχέση ε, τον Ιούνιο. Έχουμε ήδη συμφωνίες με αρκετές χώρες όπως με τη Γεωργία, τη Μολδαβία ή την Ουκρανία. Πέρα λοιπόν από την εφαρμογή των ε, μεταρρυθμίσεων, εγώ επιθυμώ να συνεργαστώ με όλους αυτούς για να εμβαθύνουμε την ε, τομεακή συνεργασία με χώρες οι οποίες είναι έτοιμες. Η Ουκρανία πάντα ε, θα έχει την ιδιαίτερη προσοχή μου γιατί έχει στρατηγική γεωγραφική θέση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα εξακολουθήσουμε να στηρίζουμε την εξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακαιρεότητα της Ουκρανίας. Ε, θα προσπαθήσουμε να τελειώσει η σύγκρουση στο Ντομπάς, να στηρίξουμε τις μεταρρυθμίσεις είτε στον τομέα κράτους δικαίου είτε στην οικονομία. Πρέπει να κάνουμε πλήρη χρήση όλων των εργαλείων μας συμπεριλαμβανομένης ε, και της υποστήριξης που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ουκρανία. Το Αζερβαϊτζάν μπορεί να είναι καθοριστικό εταίρος σε θέματα ενέργεια, αλλά πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου και το κράτο δικαίου και τη δημοκρατία. Με την Αρμενία πρέπει να εστιάσουμε στην οικονομική ανάπτυξη ανάπτυξη και με τη Λευκορωσία να βοηθήσουμε στην, στον εξυγχρονισμό της χώρας, ε, ενώ ε, να συνεχιστούν οι προσπάθειες για βασικές δημοκρατικές αξίες. Εγώ θα συνεχίσω να συνεργάζομαι για βασικά θέματα, όπως είναι το κράτος δικαίου, ο αγώνας κατά της διαφθοράς ε, και τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωση στην κοινωνία των πολιτών. Όσον αφορά τη γειτονία με την, το Νότο, βασική πρόκληση είναι η σταθερότητα, η ασφάλεια, η ευημερία και η μετανάστευση στόχοι μας θα πρέπει να είναι ρεαλιστικοί, επίσης όμως και πολύ πιο φιλόδοξοι όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή. Χάρη στην αρχή το, του περισσότερου στους περισσότερους ενθαρρύνουμε τις χώρες εταίρους μας να πετύχουν τους στόχους των μεταρρυθμίσεων. Θα θέσω σαν προτεραιότητα να προωθήσω στο πλευρό τους, στο πλευρό τους την ορθή διακυβέρνηση, την προστασία του περιβάλλοντος και προστασία του κλίματος και πιο αποτελεσματική προσέγγιση για τα θέματα τα μεταναστευτικά. Θα δώσω απόλυτη σημασία στην οικονομική ανάπτυξη και την επιτυχία των πολιτικών απασχόλησης, κυρίως όσον αφορά τους νέους. Για να πετύχουμε θα πρέπει να επικαιροποιήσουμε τις προτεραιότητες μας, να λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα συμφέροντα του καθενός από τους εταίρους μας. Το Μαρόκο, παραδείγματος χάρη, έχει μια δυναμική εξυγχρονισμού που υπόσχεται πολλά. Θα πρέπει να το υποστηρίξουμε αυτό όπως και την Τινησία και την Ιορδανία. Σε συνεργασία στενή με τον Γιώζεφ Μπορέλ έχω πρόθεση γρήγορα να υποβάλω νέες προτάσεις για τις προτεραιότητες εταιρικής σχέσεως για να αντατικοποιήσουμε τις σχέσεις μας με τις χώρες αυτές που θα πρέπει να πραγματοποιήσουν απαιτητικέ μεταρρυθμίσεις. Οι σχέση με τη Λιβύη και τη Συρία είναι πιο περίπλοκες. Η Πρώτος από τους στόχους θα είναι να εργαστώ για να ε, προωθήσω την ειρήνη και σταθερότητα σε συνεργασία με τον ΙΕ. Η σταθερότητα της Αιγύπτου εξίσου είναι ουσιώδης για όλη την περιοχή. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις οικονομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε το διάλογό μας των στενό όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Άοκνα θα εργαστούμε, συνεργαζόμενοι με μετανάστευση με τους εταίρους μας του Νότου. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για να πετύχουμε τους στόχους μας. Θα τονίσουμε βασικά την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων θα καταπολεμήσουμε επίσης κατά της παράτυπης μετανάστευσης, κατά το εμπορίου των ανθρωπίνων όντων και του παράνομου, παράνομης κυκλοφορίας των μεταναστών. Θέλουμε να αυξήσουμε την ασφάλεια και τον έχω των συνόρων, να τονώσουμε το μηχανισμό επανεισδοχή και των επιστροφών. Θέλουμε να προωθήσουμε καλύτερα την κινητικότητα και την νόμιμη μετανάστευση. Ε, αυτό θα είναι κάτι υποφέλε και τι δύο πλευρές. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε το Λίβανο και την Ιορδανία, δύο χώρες που θα έχουν υποδεχτεί πολύ μεγάλο αριθμό προσφύγων. Θα πρέπει τέλος να υποστηρίξουμε την εθελοντική επιστροφή στη Συρία εάν οι βασικές οι βασικοί όροι για αξιοπρεπή και ασφαλή επιστροφή των μεταναστών και των προσφύγων γίνονται σεβαστέ ε, σε στενή συνεργασία με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Αξιότιμα μέλη. Για να υποστηρίξουμε τους στόχου θα ήθελα λοιπόν να μου επιτρέψετε να ανακεφαλαιώσω στα τέσσερα βασικά που πρέπει να επιτύχουμε τα επόμενα χρόνια. Πρώτον, πρέπει να ανοίξουμε τι ε, διαπραγματεύσει ε, ένταξη ε, με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Και αυτό σημαίνει να του δώσουμε μια σαφή προοπτική ένταξη με βάση αρχέ που έχουμε ανακοινώσει. Επίση, πιο αποτελεσματική διαδικασία να προετοιμαστούμε για να επιτύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα στου στην καθημερινή του ζωή. Άρα δηλαδή να στηρίξουμε τις μεταρρυθμίσεις, να αυξηθεί ουσιαστικά ε, η οικονομική και χρηματοδοτική μας υποστήριξη με στόχο να βελτιωθεί η οικονομία, το εμπόριο, η εκπαίδευση και οι συνθήκες ταξιδιών. Δεύτερον, οι χώρες ε, της ανατολικής συνεργασίας ε, θα πρέπει να βελτιώσουν την οικονομία τους, τη σταθερότητα. Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την εδαφική καιρότητα της Ουκρανίας, να τη στηρίξουμε στην αντίστασή της. Τρίτον, θα ανανεώσουμε τη συνεργασία μας ε, με την ε, νότια γειτονική συνεργασία. Θα βοηθήσουμε στην οικονομική ανάπτυξη των εταίρων. Τέταρτον, θα κάνουμε πλήρη χρήση του εργαλείου της ε, γειτονική σχέσης και επίσης και του εργαλείου του προενταξιακού. Με τον τρόπο αυτό θα εστιάσουμε περισσότερο στις επενδύσεις. Επίσης θα στηρίξουμε τη συνεργασία με τους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς για να έχουμε καλύτερες μεταρρυθμίσεις. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, εάν τελικά με επιβεβαιώστε στη θέση του Επιτρόπου, εγώ θα αναζητήσω την συνεχή και στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Θα συνεργάζομαι στενά με αυτήν και άλλες επιτροπές. Θα υπάρχει άμεση σχέση ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, ε, και τους εταίρους μας ε, και ε, θέλω να μπορώ να βασιστώ πλήρως στην διπλωματική δύναμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πρέπει να μιλάμε με μία φωνή, να βασιζόμαστε σε κοινέ αρχές. Εγώ θα είμαι στη διάθεση διάθεσή σας για ε, συζητήσεις ε, για τη δουλειά μας και ειλικρινά ελπίζω ότι αυτή η ακρόαση ε, θα δρομολογήσει μια ανοιχτή και επικοδομητική συνεργασία. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε κύριε υποψήφιε επίτροπε. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για τις ε, εισαγωγικές σας παρατηρήσεις και τώρα περνάμε στον πρώτο γύρο των ερωτήσεων και Πρώτο ομιλητή εκ μέρου του ΕΛΚΟ, ο κύριο Ζαβνόφκοβ, για ένα λεπτό. Η κυρία, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ. Η υπερό μα έχει γίνει ειρηνική και πιο πλούσια χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συνεργασία. Ωστόσο, η πορεία των Δυτικών Βαλκανίων εμποδίζεται λόγω εχθρότητας που υπάρχει μεταξύ των χωρών. Είναι σημαντικό να υπάρξουν πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις και να υποστηριχθούν τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων στην ε, πορεία τους προς την εκπλήρωση των κριτηρίων της Κοπενχάγης. Έχοντας αυτό κατά νου, πώς μπορούμε να επιταχύνουμε την ένταξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, ιδίως στους δύσκολους τομείς της επανασυμφιλίωσης, της δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η περιφερειακή συνεργασία σε μια περιοχή που είναι δύσκολη ε, δείχνει ότι πρέπει πολλά να γίνουν ακόμη ε, ιδίως στον τομέα της συμφιλίωσης. Ποια θα είναι τα συγκεκριμένα μέτρα που θα λάβετε για να προωθήσετε την περιφερειακή συνεργασία στα Δυτικά Βαλκάνια. Κύριε Υποψήφιο Επίτροπε, παρακαλώ, δύο λεπτά έχετε στη διάθεση σας. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να υπογραμμίσω σαφώς ότι παρά το γεγονός ότι υπήρξαν κάποιες δυσκολίες, αν θέλετε, ε, στην Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου, Κανείς, μα κανείς, ούτε σε εκείνη τη συζήτηση που έγινε τον Οκτώβριο, δεν αμφισβήτησε την προσήλωση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ε, τελική ένταξη των ε, Δυτικών Βαλκανίων. Αυτό δεν έχει αλλάξει και εγώ θα αγωνιστώ μέχρι τέλους για να υλοποιηθεί αυτός ο στόχος. Βεβαίω θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι πρέπει και να ενισχύσουμε την δουλειά μας γιατί εκφράστηκαν ανησυχίες οι οποίες πρέπει να γίνουν σεβαστές και να αντιμετωπιστούν. Εγώ εκφράζω την προθυμία μου και την πρόθεσή μου να συνεργαστώ με τις χώρες που εξέφρασαν τις ανησυχίες καθώς και με τις χώρες που καλούνται να τις αντιμετωπίσουν. Στη συζήτηση αυτή είναι βασικό ζήτημα το κράτος δικαίου και στον τομέα τη ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη και τη διαφορά πρέπει να ενισχύσουμε τη συνεργασία μα με τα Δυτικά Βαλκάνια. Από την άλλη πλευρά πρέπει να ανταποκριθούμε και εμεί στι δεσμεύσει μα. Δηλαδή, να γίνει πραγματικότητα η προσχώρηση των, χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θεωρώ ότι μία από τι μεγαλύτερε προκλήσει είναι το μεγάλο χάσμα που υπάρχει όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη ανάμεσα σε εκείνες τις χώρες και σε εμάς. Και εγώ θα κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου στη διάρκεια των πέντε αυτών ετών, αν επιβεβαιώσετε την υποψηφιότητά μου, να κλείσει το χάσμα αυτό και να φέρω οικονομική ευημερία και ανάπτυξη στις χώρες αυτές. Και βεβαίως είναι δεδομένο ότι η οικονομία της αγοράς δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς το κράτος δικαίου. Αυτά τα δύο συμβαδίζουν. Για την περιφερική συνεργασία θα επιδιώξω να ενισχύσω τις σχέσεις μεταξύ των χωρών αυτών με ουσιώδη τρόπο, διότι διαφορετικά δεν θα μπορέσουν ποτέ να διαδραματίσουν το ρόλο που πρέπει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Κυρία Ζόφκο, θέλετε να κάνετε κάποια συμπληρωματική ερώτηση. Η κατάσταση Βοσνία Ροζεγοβίνη είναι περίπλοκη και η χώρα αυτή είναι εκτεθειμένη και σε δράσεις ε, παραγόντων εκτός ε, Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Ποια είναι η γνώμη σας για τη στάση του ΟΗΕ και του ειδικού απεσταλμένου στην περιοχή. Ποια είναι η δική σας ε, πρόθεση ώστε να ε, εδρεωθεί η σταθερότητα και η ειρήνη στην περιοχή και ποια είναι η άποψή σας για την Βοσνία Ερζεγοβίνη, ποια είναι δε τα διδάγματα που, έχουμε αντλήσει, που έχετε αντλήσει από το παρελθόν. Ευχαριστώ κύριε υποψήφιο επίτροπε, έχετε ένα λεπτό και από εδώ και πέρα θα είμαι πιο αυστηρός με το χρόνο σας. Το κλειδί στις σχέσεις μας με τη Βοσνία Ζεγοβίνη είναι η εφαρμογή των 14 σημείων που έχει αναλύσει και συντάξει, προσδιορίσει η Κομισιόν ως τομής προτεραιότητας για τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν στη χώρα. Πρέπει να συνεργαστούμε με τη Βεσνία ε, Ερζεγοβίνη, με την κυβέρνηση της χώρας αυτής, την οποία δεν έχει η χώρα εδώ και ένα χρόνο και καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί μια χώρα να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν έχει κυβέρνηση και δεν υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσει που πρέπει. Εμεί θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μα για να του βοηθήσουμε. Για την ε, δραστηριότητα και τη συμμετοχή των, ε, των Ηνωμένων Πολιτειών ε, εγώ εκφράζω την πρόθεσή μου να συνεργαστούμε στενότατα για, την, για τα θέματα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης. Κύριε υποψήφιο, κύριε υποψήφιο επίτροπε, κύριε Βαρχένη, η Ευρωπαϊκή Επίτροφη είναι εκτελεστική εκπρόσωπη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να υπερασπίζονται τις κοινέ μας αξίες. Κατέρχεται της θητεία σας, σαν μόνιμος εκπρόσωπος της Ουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είσαστε εκείνο που έχετε να παρουσιάσετε και να υπερασπιστείτε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τις μεταρρυθμίσεις της Ουγγρικής Κυβερνήσεως. Κάποια νομοσχέδια που θέτει η Ουγγαρία παραβίαζαν σαφώ τι συνθήκε. τη χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων και τα κριτήρια της Σαν αποτέλεσμα, η διαδικασία του άρθρου 7 τη συνθήκη Ευρωπαϊκή Ενώσεω που ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο ξεκίνησε κατά τη Ουγγαρίας σαν επίτροπος για διεύρυνση. Πώ θα εξασφαλίζεται ότι στις υποψήφιε χώρε το κράτο δικαίου ακρογωνίω λίθο των κριτηρίων τη Κοπενχάγη και αξία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω θα εφαρμόζεται στην ουγγρική πολιτική εσείς ε, πολύ συχνά ε, περασπιζόσατε την αντίθετη θέση. Κύριε Βερχέη, δύο λεπτά έχετε το χρόνο να απαντήσετε. Σαν επίτροπος καθήκον μου θα είναι να εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό θα κάνω. Όπως θα είδατε, στα προηγούμενά μου καθήκοντα ήδη εργαζόμουν ανεξάρτητα από οδηγίε κυβερνήσεων σαν δημόσιος υπάλληλο Ευρωπαίος. Προτίθεμαι να κάνω το ίδιο και να ακολουθήσω την ίδια προσέγγιση εργαζόμενος ως Ευρωπαίος Επίτροπος ακολουθώντας τη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και μόνο τη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Όσον αφορά το κάτος δικαίου στα Δυτικά Βαλκάνια, Έχουμε σαφέστατα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται και δεν προτίθεμαι να αλλάξω ή να προτείνω η αδίποτε αλλαγή στα εν λόγω κριτήρια. Αντιθέτως, όπως εξήγησα στην προηγούμενη απάντηση, πιστεύω ότι πρέπει να εντατικοποιήσουμε τη συνεργασία με τους γείτονές μας Δυτικών Βαλκανίων να πετύχουμε περισσότερα, διότι ήταν ένας από τους λόγους αυτό για τον οποίο τρία κράτη-μέλη εξέφρασαν σημαντικές ανησυχίες τον τελευταίο χρόνο. Θα επεξεργαστώ, επεξεργαστώ αυτούς τους τομείς σαν τομεί προτεραιότητας σε συνεργασία με αυτέ τι χώρες και με τα ενδιαφερόμενα προαναφερθέντα κράτη-μέλη. Νίνο Πίτσουλα, συμπληρωματική ερώτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ποια συγκεκριμένα βήματα θα λάβετε αν η αδίποτε χώρα διεύρυνσης υιοθετήσει μέτρα που δεν συνάδουν με τι βασικέ αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω, κυρίως όσον αφορά τη δημοκρατία, το κάτω δικαίου, συμπεριλαμβανομένης ανεξαρτησία του δικαστικού κλάδου και της καταπολέμησης διαφθορά. Στη γραπτή απάντηση στη δεύτερη ερώτηση αναφέρατε ότι προσδίδεται μεγάλη σημασία στην ισότιμη αντιμετώπιση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στα πλαίσια των δημοσιονομικών μέσων. Θα ήθελα να ξέρω, αναλαμβάνετε την υποστήριξη την δημοκρατική αιρεσιμότητα που επιτρέπει την ανεξαρτησία των διαφόρων φορέων και μπορείτε να επικαιροποιήσετε όλα τα παρατήματα ενταξιακών συμφωνιών. Υποψήφια Επίτροπε. Αρχή μας, στα Δυτικά Βαλκάνια, είναι η αρχή που εκπροσωπείται και αντιπροσωπεύεται την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι τα θεμελιώδη πρέπει να πηγαίνουν πρώτα. Και αυτό θα επιδιώξω. Τι σημαίνει αυτό. Ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει πρόοδο όσον αφορά το κράτο δικαίου, δεν μπορεί να υπάρχει πραγματική πρόοδο στην ενταξιακή διαδικασία. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω κάθε μέσο διαθέσιμο για να εξασφαλίσω ότι το κράτος δικαίου και η ρεσιμότητα όσον αφορά το κράτος δικαίου θα είναι κάτι που θα σέβονται οι γειτονέ μα και τέροι μα. Εάν δεν ισχύει κάτι τέτοιο, θα πρέπει να ακολουθήσω σταδιακή προσέγγιση που ίσως να οδηγήσει και σε αναστολή της χρηματοδότησης. Όσον αφορά του δημοσιονομικούς κανονισμούς για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, αυτό είναι κάτι που θα συζητήσουμε στο μέλλον. Οι αρχές που ακολουθώ σύμφωνα με αυτό είναι ότι θέλουμε να έχουμε μέσα οικονομικά που είναι διαθέσιμα, πραγματιστικά, αποτελεσματικά και ευέλικτα. Ε, βεβαίως θα πρέπει να εξετάσουμε τη διαχείριση αυτών και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα λαμβάνονται υπόψη. Και τώρα το λόγο έχει η ομάδα Renew, ο κύριος Κούτσοκ. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, σας καλωσορίζουμε στην Επιτροπή μας, στη συνάντησή μας. Μας παρουσιάσατε έτσι μια πολύ μεγάλη εικόνα για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απέτυχε στο να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Εγώ δεν βλέπω τι μπορεί να γίνει στα Δυτικά Βαλκάνια. Πριν από πέντε χρόνια ο κύριος Γιούγκερ είπε νομίζω τότε στο Στρασβούργο ότι για τα επόμενα πέντε χρόνια δεν θα υπάρξει διεύθυνση. Μεγάλο το λάθος του τότε, αλλά εν πάση περιπτώσει ανήκει στο παρελθόν. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πεπισμένο ότι πρέπει να υπάρξει διεύρυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ίδιο ισχύει και για την Επιτροπή. Πρόβλημα είναι το Συμβούλιο. Εσείς λοιπόν πώς θα μπορέσετε να το πείσετε. Τώρα, η δεύτερη ερώτησή μου είναι ένα μεγάλο δίλημα, δηλαδή ανάμεσα στην εμβάθυνση και τη διεύρυνση. Ποια ακριβώ ε, είναι η άποψή σας που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρώτα να γίνουν εσωτερικές αλλαγές και ε, να υπάρξουν τέτοιου είδους εξελίξεις πριν ξεκινήσουν οι προενταξιακές ε, διαργασίες. Και τελικά, ε, εάν ξεκινάνε προενταξιακές διαπραγματεύσεις, ποιες θα πρέπει να είναι οι προϋποθέσεις. Ο κύριος υποψήφιος, παρακαλώ, για δύο λεπτά. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά στην προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Θέλω να υπογραμμίσω ότι Ακόμα και αν δεν κατορθώσαμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου, υπάρχει παρόλα αυτά πλήρης δέσμευση και του Συμβουλίου όσον αφορά τις προοπτικές αυτών των δύο κρατών. Και η δική μου πρόθεση είναι να άρω όλα τα εμπόδια που υπάρχουν και φάνηκαν στη συζητήση στο Συμβούλιο. Θα τίνω χειραβοητεία σε αυτές τις χώρες και από την πρώτη και όλες μέρα που θα αναλάβω, αν τελικά με επιβεβαιώσετε στη θέση μου, θα προσπαθήσω να δω ε, τις συγκεκριμένες εξελίξεις. Νομίζω ότι εδώ υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας είναι να διασφαλίσουμε ότι η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία θα έχουν τελικά διαπραγματεύσει, διαπραγματεύσεις, ενταξιακέ, πριν από τη συνάντηση κορυφή στο Ζάγκρεπ. Και πρέπει να εργαστούμε ε, πάνω στις ανησυχίε που έχουν κυρίω σχέση με το άσυλο, ε, ψεύτικες ε, τη ασύλου που έχουν σχέση με τη διαφθορά και κάποια άλλα στοιχεία της ευνομία. θα ασχοληθώ με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία για να φύγουν αυτές οι ανησυχίες, να ε, εξοβελιστούν και για να καλύπτονται τα κριτήρια. Όσον αφορά τώρα σε αυτήν την νέα Επιτροπή που θα προκύψει, νομίζω ότι υπάρχει ένα σαφέστατο μήνυμα από την υποψήφια πρόεδρο ε, σχετικά με το ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή προοπτική αυτών των κρατών. Αυτό που ρωτήσατε για το δίλημα μεταξύ διεύρυνση και εμβάθυνση, εγώ δεν πιστεύω ότι το ένα αποκλείει το άλλο πρέπει να προσπαθήσουμε έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει πιο αποτελεσματική, πιο ισχυρή, αλλά αυτό που δεν, είναι, δεν μας εμποδίζει στο να προχωρήσουμε και στον δρόμο της διεύρυνσης. Ευχαριστούμε πολύ. πολύ συντομή συμπληρωματική ερώτηση όσον αφορά το πλαίσιο. Γιατί νομίζω ότι αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο. Εσείς, χρονικό πλαίσιο, πώς το βλέπετε αυτό σχετικά με την αναθεώρηση αυτής της διαδικασίας μέχρι να προκύψει μια νέα μέθοδος. Ο κύριος Βαχαή, για ένα λεπτό παρακαλώ. Εγώ δεν νομίζω ότι το θέμα του πλαισίου της διεύρυνσης, το σύνολο του, ότι πρέπει αυτό να αναθεωρηθεί. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να ενισχυθεί η μέθοδος και μάλιστα με ένα τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να προκύψει μεγαλύτερος δυναμισμός, περισσότερες δυνατότητες αυτές οι υποψήφιες χώρες να αναπτύξουν δυναμισμό. Οι χώρες αυτές που μπορούν και επιθυμούν να εξελιχθούν με μεγαλύτερη ταχύτητα αφενός και αφετέρου για τις άλλες που ε, θα προχωράνε με ε, αργότερο ρυθμό και εκεί πρέπει να είναι πιο αργή η όλη διαδικασία της διεύρυνσης. Έχουμε διαπιστώσει ότι οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να καλύπτονται πριν ε, από όλα υπάρχουν αυτές οι βασικές προϋποθέσεις και νομίζω πρέπει να είμαστε απόλυτα σαφείς ότι οι προϋποθέσεις αυτές θα παραμείνουν ακριβώς οι ίδιες. Ευχαριστώ. Εκ μέρους των ε, Πρασίνων το λόγο έχει ο κύριος Έρνεστ Ουρτασούν. Ευχαριστώ κύριε Υποψήφιο Επίτροπο που είστε εδώ. Είστε πάντα ήσασταν πάντοτε υπέρμαχος των προτεραιοτήτων του κυρίου Όρμπαν εδώ στις Βρυξέλλες και ταυτόχρονα ο κύριος Όρμπαν θεωρεί ότι το χαρτοφυλάκιο αυτό είναι εθνικό του περισσοϊκό στοιχείο. Και αυτό ε, ήταν σαφές και στην Σύνοδο Κορυφής του Συμβουλίου όπου ε, υποσχέθηκε ε, στενή συνεργασία με την Τουρκία αν η κυβέρνηση του πάρει το χαρτοφυλάκιο, αλλά υποσχέθηκε κιόλας ότι θα ανταποκριθεί στις ελπίδες του. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα αφοσίωσης. Πρέπει εσείς να μας ε, αποδείξετε ότι θα είστε αφοσιωμένος στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Και αυτά είναι πολύ ανησυχητικά. Θέλω λοιπόν να σας δώσω τώρα την ευκαιρία να μας δείξετε την αφοσίωσή σας. Ε, καταδικάζοντας ή παίρνοντα αποστάσεις από αυτήν την δήλωση του κυρίου Όρμπαν. Γιατί θα είναι πολύ ανησυχητικό ε, αν δεν το πράξετε. Είστε ε, έτοιμος να δηλώσετε τη διαφωνία σας με, τα, με τις δηλώσεις του κυρίου Όρμπαν. Ο κύριος Βαρέλη. Από την ημέρα που θα αναλάβω τα καθήκοντά μου, εγώ ως Επίτροπος θα είμαι πλήρως ανεξάρτητος, δεν θα παίρνω καμία οδηγία από καμία κυβέρνηση, από κανένα θεσμικό έργο. Θα είμαι μέλος του Σώματος των Επιτρόπων. Με συναδελφικό τρόπο λοιπόν θα υπερασπίζομαι και θα εφαρμόζω την ευρωπαϊκή γραμμή και μόνο. Ευχαριστούμε. Κύριε Ουρτασούν, θέλετε να κάνετε κάποια συμπληρωματική ερώτηση. Ναι, όπως φαντάζεστε, φαντάζεστε αυτό δεν μας αρκεί. Ωραία ήταν τα λόγια αυτά, αλλά είμαστε εδώ όπου μια εθνική πρωτεύουσα παρεμβαίνει στο χαρτοφυλάκιό σας λέγοντάς σας τι, έχετε, τι πρέπει να κάνετε. Αυτό είναι απαράδεκτο για επίτροπο. Είναι ανησυχητικό και πρέπει πραγματικά να ε, καταδικάσετε αυτήν την στάση. Γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσετε να εφαρμόσετε ευρωπαϊκή πολιτική. Δεν γίνεται αυτό με ωραία λόγια. Πρέπει ενεργά να σταθείτε αντίθετα προς την ε, πρόθεση την εκπεφρασμένη πρωτεύουσα να επηρεάσει το έργο σας ως Επιτρόπου. Κύριε Επιψήφιε Επίτροπε, εγώ ως Επίτροπος δεν θα ε, δεχτώ καμία παρεμβολή, καμία παρέμβαση όσον αφορά την άσκηση των καθηκόντων μου από καμία κυβέρνηση, από καμία πρωτεύουσα. Ευχαριστώ. Ομάδα ID. Η κυρία Άννα Μπονφρίσκο έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κύριε Επίτροπε. Καλώς ήρθατε υποψήφια Επίτροπε. Μιλάω Ιταλικά. Στα Ιταλικά γιατί θέλω να εμβαθύνουμε στο θέμα της Μεσογείου. Εσείς πριν, πριν αναφερθήκατε σε κάποιες βασικές σημαντικές χώρες. Η ερώτηση είναι κατά την άποψή σας ποιον ακριβώς ρόλο θα πρέπει να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές τις χώρες της νότιας ακτής της Μεσογείου για να προωθήσει αλλά και για να πετύχει μια πραγματική πολιτική δημοκρατική σταθερότητα, οικονομική σταθερότητα, να πετύχει ασφάλεια που θα επιτρέπει σε μας να βλέπουμε με αισιοδοξία μια διαδικασία διαλόγου Ευχαριστώ κυρία μου. Ο κύριος Βεχέια, δύο λεπτά. Στη νότια γειτονιά, στη νότια γειτονία μας, λαμβάνω υπόψη σαν παράδειγμα το Μαρόκο. Το Μαρόκο είναι πρόθυμο να συνομιλεί μαζί μας και να συνεργάζεται όχι μόνο σε τομείς που ενδιαφέρουν το Μαρόκο, αλλά και που συμφέρουν και ενδιαφέρουν εμάς. Γι' αυτό μπορούμε να συνεχίσουμε αναπτύσσοντας περαιτέρω αυτή τη συνεργασία μαζί τους συνεργάζονται μαζί μας στη μετανάστευση. Αυτό το θεωρώ σημαντικότατο για τα συμφέροντά μας. Θα πρέπει να συνεργαστούμε καλύτερα για οικονομική ανάπτυξη, ξένες άμεσες επενδύσεις και ακόμα εμπόριο. Και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει μοντέλο πρότυπο για όλη τη νότια γειτονιά. Βλέπω πολλές δυνατότητες και σε σχέση με την Τινησία, από τη στιγμή που θα έχει καινούρια κυβέρνηση, θα έχουμε νέο πρόεδρο στον Σαχίτ που θα μπορούσε να είναι εταίρος μας σε μια τέτοια προσπάθεια. Έτσι θα μπορούσαμε να αυξήσουμε τις δυνατότητες οι λαοί αυτών των χωρών αυξάν δυνατότητες αυτοί οι λαοί να έχουν δουλειά, να βρουν δουλειά και μια ζωή με νόημα στις πατρίδες τους. Αυτό επίσης σημαίνει βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος, ε, βελτίωση της δημόσιας δίκησης. Μπορούμε να συμβάλλουμε πάρα πολύ στις προσπάθειες της περιοχής. Αυτοί θα πρέπει να συνεργαστούν μαζί μας σε τομείς όμως που είναι και ύψη σημασίας για μας. Ευχαριστώ. Κύριε Μαφρίσκο, ε, συμπληρωματική ερώτηση. Λοιπόν, ποιες είναι οι προτεραιότητες πέρα από τις χώρες που αναφέρατε και συμφωνώ με την άποψή σας, αλλά οι προτεραιότητες που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίσει στη Λιβύη, παραδείγματος χάρη, ή στο Λίβανο, ή και στην ίδια την Ένωση για τη Μεσόγειο, για να επαναπροωθηθεί η δράση εκεί της Ευρωπαϊκής Ενώσεως που δεν έδωσε ε, μεγάλα αποτελέσματα, μέχρι τώρα τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ. Κύριε Βερχέη. Στη Λιβύη αντιμετωπίζουμε δύο προβλήματα το πρώτο είναι ανθρωπιστικό, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει και θα έπρεπε να βοηθήσει και πρέπει να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας για να βελτιώσουμε τις ε, συνθήκες για τους μετανάστες ανθρωπιστικές, να βοηθήσουμε την κυβέρνηση να εξασφαλίζει συνθήκες που να είναι στο ύψος των δικών μας προτύπων και προδιαγραφών όσον αφορά τους ε, πρόσφυγες. Από την άλλη πλευρά, η χώρα ε, έχει έναν εμφύλιο πόλεμο πρέπει να σταθεροποιηθεί. Αλλά εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να κινηθεί μόνη τη. Χρειαζόμαστε του άλλου εταίρου μα στον κόσμο να μα βοηθήσουν να σταθεροποιήσουμε την ε, χώρα. Λοιπόν, θα πρέπει να συμμετάσχουν οι Ηνωμένε Πολιτείε, ούτω ώστε να μα βοηθήσουν να φέρουμε την ειρήνη στη χώρα. Για το Λίβανο. Το ο Λίβανο φιλοξενεί ένα από του μεγαλύτερου πληθυσμού προσφύγων. Συνεργαζόμαστε ίδιο με το Λίβανο πρέπει να ανταδικοποιήσουμε και εκεί τις προσπάθειές μας, να τους βοηθήσουμε να φροντίσουν για όλους αυτούς τους πρόσφυγες. Από την άλλη πλευρά βέβαια, η οικονομική ανάπτυξη, οι δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης υπάρχουν στο Λίβανο, όμως η κατάσταση της ασφαλείας πρέπει να σταθεροποιηθεί σε αυτή τη χώρα. Η Άννα Φωτίγκα για το ECR. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε υποψήφιε. Επίτροπε, σας καλωσορίζουμε στην Επιτροπή μας. Ε, ο κύριος Γιούγκερ πριν από πέντε χρόνια ε, μίλησε για τη διεύρυνση και επίσης ε, και είχαμε και πρόσφατες αποφάσεις που αφορούν στη Βόρεια Μακεδονία και στην Αλβανία. Και αυτά επηρέασαν ουσιαστικά τις χώρες που εντάσσονται στη διαδικασία της Θεσσαλονίκης, επηρέασαν όμως και τις χώρες της ανατολικής εταιρικής σχέσης. Με αυτές τις χώρες πρέπει να βρούμε έναν τρόπο έτσι ώστε να ε, ανανεώσουμε την, ε, το ενδιαφέρον τους ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίως ε, θα πρέπει να επαναφέρουμε τις σχέσεις με τις χώρες Ουκρανία, Γεωργία, Μολδαβία που είναι συνδεμένες με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και με άλλες χώρες. Ποια είναι τα δικά σας τα προγράμματα. Ευχαριστούμε κυρία Φωτίγκα. Κύριε υποψήφια έχετε δύο λεπτά. Αυτή τη στιγμή ε, αναθεωρούμε την ε, ανατολική εταιρική σχέση. Μέχρι τώρα, τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να σκεφτεί το τι θα προτείνει για το μέλλον της ε, ανατολικής εταιρικής σχέσης. Η δική μου άποψη σχετικά με την ε, ενίσχυση της ανατολικής εταιρικής σχέσης είναι να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές να αποκτήσουν μια οικονομία της αγοράς η οποία ε, θα τις βοηθήσει να αντισταθούν σε εξωτερικές πιέσεις αλλά και επίσης να δημιουργηθεί ένα κλίμα επενδύσεων το οποίο θα είναι προς όφελος αυτών των κρατών. Όσον αφορά τώρα στις, ε, σε εκείνες τις χώρες της ανατολικής εταιρική σχέσης, Εάν οι χώρες αυτές ε, θέλουν να συνεργαστούν περισσότερο μαζί μας, καλώς έχει να ενταχθούν ε, σε όσο περισσότερους τομείς επιθυμούν. Από την άλλη βέβαια πρέπει να υπογραμμίσω ότι τα εργαλεία αυτά και οι προποθέσεις αυτές ε, πρέπει να εφαρμοστούν γιατί οι χώρες αυτές ε, ανέλαβαν να εφαρμόσουν περίπου το 70% της αρμοθεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να τις βοηθήσουμε λοιπόν ως εκ τούτου Υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να ολοποιηθούν σχετικά με τις ε, προϋποθέσεις που ισχύουν, αλλά να γίνουν και πολλά περισσότερα όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, βασικές υποδομές, όπως είναι οι μεταφορές, η ενέργεια, αλλά και όσον αφορά ναι. τις ε, πράσινες συμφωνίες ε, θα πρέπει να συνεργαστούμε περισσότερο με αυτές τις χώρες όσον αφορά τις συνολικές συμφωνίες ελεύθερων εμπορικών ανταλλαγών, τα περίφημα EDFTAs. Θέλω να σας ρωτήσω το εξή. Ε, υπάρχει κάποιο περιθώριο συνεργασίας ε, και με τις χώρες ανατολικής ε, εταιρικής σχέσης, αλλά κάποιες εξ αυτών, η Λευκορωσία παραδείγματο χάρη, εκεί υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Γιατί στη Λευκορωσία γίνονται πράγματα που στρέφονται εναντίον μας. Αλλά υπάρχουν άλλες χώρες όπως ας πούμε η Ουκρανία, η οποία ε, Ουκρανία αγωνίζεται κατά της εξωτερικής ε, επιθετικότητας και σε κάποιο βαθμό αγωνίζονται εξ ονόματος όλων μας. Οι συνδεδεμένες χώρες έχουν συμφωνίες πλαίσιο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Παραδείγματο χάρη η ε, Ουκρανία έχει ε, συνάψει μία συμφωνία που αφορά στα θέματα της ε, διοίκησης. Ο κύριος Επίτροπος έχει το λόγο. Όπως σας είπα και προηγουμένως, εάν θέλουν οι χώρες αυτές να συνεργαστούν περισσότερο μαζί μας, και σε θέματα ασφάλειας, βεβαίως και θα το κάνουμε. Όσον αφορά στην Ουκρανία, έχουμε ειδική ευθύνη για τη χώρα αυτή πρέπει να τη βοηθήσουμε να ανακτήσει την κυριαρχία της ε, στο σύνολο του εδάφους της Ουκρανίας και πρέπει να τη στηρίξουμε την Ουκρανία για να μην ε, συνεχίζονται οι κυρώσεις ε, έναντι της Ρωσίας όσο δεν υπάρχει πρόοδο στη διαδικασία μην θα συνεχίσουν να ισχύουν οι κυρώσει. Εγώ βέβαια δεν έχω τα εργαλεία που έχει ο κύριος Μπορέλ στο δικό μου το χαρτοφυλάκιο, όμως εγώ θα στηρίξω όλες τις ενέργειες για να βοηθήσουμε την Ουκρανία να ανακτήσει την κυριαρχία της. Πάμε τώρα στην επόμενη ομάδα, στο, το λόγο στον κύριο Γεωργίου. Επίτροπε, ενώ μιλάτε για την ανάγκη οικοδόμησης ενός κράτους δικαίου στα Δυτικά Βαλκάνια. Η χώρα σας, ο Πρωθυπουργό σας, αλλά και εσείς, ως μόνιμος αντιπρόσωπος της Ουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εγκαλείστε και μέσα από την ενεργοποίηση του άρθρου 7 της συνθήκης της Λισαβόνας. Ε, είστε υπόλογοι για την υπόσκαψη κάποιων θεμελιωδών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερώτηση τελικά θα είστε ένας διχασμένος επίτροπος και θα πατάτε σε δύο βάρκες. Η μια θα είναι η ψυχή σας και αυτό που πραγματικά πιστεύετε και το άλλο θα είναι η ανάγκη να εξυπηρετήσετε τη θέση στην οποία θα διοριστείτε, αν διοριστείτε. Thank you, Ευχαριστώ συνάδελφε, κύριε υποψήφιο επίτροπε. Έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή σας. Ως επίτροπος, εγώ θα επιδιώξω την εφαρμογή των θέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά το κράτος δικαίου, είτε στα Δυτικά Βαλκάνια, είτε στην Ανατολική Εταιρική Σχέση, είτε στην Νότια Γειτονία. Θα υπερασπιστώ αυτή τη γραμμή με ανεξάρτητο τρόπο, χωρίς κανένα εμπόδιο από εξωτερικές παρεμβάσεις και πάντοτε σε σύμπνοια με τους συναδέλφους μου στο Σώμα των Επιτρόπων. Συμπληρωματική ερώτηση. Ε, είναι ένα σημαντικό εταίρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια στιγμή όμω κάνατε παραδοχή ότι παραβιάζει τι αρχέ του διεθνού δικαίου και δεν πρέπει να κάνουμε τα στραβά μάτια. Ο κύριο Όρπαν όταν επικρότησε την εισβολή τη Τουρκίας στη Συρία έκανε τα στραβά μάτια. Αυτή τη δήλωση εσεί την απορρίπτετε ως δήλωση η οποία έπρεπε να γίνει γιατί δεν έπρεπε να έρθουν πρόσφυγες στην Ευρώπη. Αυτή είναι μια αντίληψη που θα βοηθήσει για την πολιτική τη διεύρυνση και για την οικοδόμηση κράτου δικαίου και για τι χώρε οι οποίε είναι υποένταξη. Κύριε υποψήφιο επίτροπε, ένα λεπτό έχετε στη διάθεσή σας. Όσον αφορά την Τουρκία, έχουμε μια ξεκάθαρη άποψη και γραμμή για το τι πρέπει να γίνει όσον αφορά το κράτος δικαίου. Εν τούτης, έχουμε δει ότι υπάρχει, έχει υπάρξει κάποια ε, υπαναχώρηση στον τομέα αυτό και αυτό είναι ο βασικό λόγο για τον οποίο έχουν τελματώσει οι προενταξιακέ διαπραγματεύσει. Θα πρέπει να γίνει σε βάθο αξιολόγηση τη μελλοντική μα σχέση με την Τουρκία. Έχουμε συμφέροντα όσον αφορά την Τελωνιακή Ένωση και τη μετανάστευση. Βεβαίω έχουμε και συγκεκριμένε ανησυχίε. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να διεξάγουν μια ει συζήτηση για το ποια θα πρέπει να είναι η μορφή των μελλοντικών μα σχέσεων με την Τουρκία όσον αφορά τι παράνομε γεωτρήσει γύρω από την Κύπρο. Οι Υπουργοί Εξωτερικών ήταν σαφείς όσον αφορά την ε, πιθανότητα επιβολή περιοριστικών μέτρων. Αν κάτι τέτοιο κρυθεί αναγκαίο, θα επιβληθούν αυτά τα περιοριστικά μέτρα. Ευχαριστώ συνάδελφοι. στον πρώτο ο πρώτος γύρο των ερωτήσεων. Από τους ομιλητές, οι συντονιστέ των ομάδων μου, στο δεύτερο γύρο, ξανά από το ΕΛΚ. Ο κ. Άντριο Καβίλιο έχει το λόγο. Κύριε υποψήφιε Επίτροπε, η Ursula Βαντερλάιν, η πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είπε ότι η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι γεωπολιτική Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στη δήλωσή σα επίση τονίσατε ότι η Ουκρανία είναι πολύ σημαντική γεωπολιτικά για σας. Συμφωνώ μαζί σας λοιπόν ότι στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο η γεωπολιτική επικεντρώνεται στην περιοχή τη Ανατολική Γειτονία. Και η κατάσταση αυτή Τρει χώρε η Ουκρανία, η Γεωργία και η Μολδαβία θέλουν να ενταχθούν, το Κρεμλίνο αντιτάσσεται και υπόσχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ένταξή τους. Στην αποστολή σας δηλώνετε ότι πρέπει να δημιουργήσετε νέους στόχους μακροπρόθεσμης πολιτικής μέχρι τα μέσα του 2020 για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική γειτονίας. Ποιοι πρέπει να είναι μακροπρόθεσμοι στόχοι για τις χώρες της Ανατολικής και ποιοι γεωπολιτικοί στόχοι θέλετε να επιτευχθούν με αυτές τις χώρες που είναι κρίσιμης γεωπολιτικής σημασίας για σας. Κύριε Βερχέ. Η πλήρη ένταξη τη Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που ζητάει η Ουκρανία θα πρέπει να το αναλύσουμε το θέμα και εμείς και να το εξετάσουμε. Μέχρι τώρα δεν έχουμε προσφέρει αυτή τη δυνατότητα στην Ουκρανία. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, ακόμα και σε αυτό το πλαίσιο, πέρα από την εφαρμογή και επιτάχυνση της εφαρμογής της συμφωνίας, της προεντεξιακής συμφωνίας με την Ουκρανία, να τους βοηθήσουμε να δημιουργήσουν μια στέρεη οικονομία της αγοράς που προσελκύει ξένες άμεσες επενδύσεις, που δημιουργεί ανάπτυξη και θέσεις εργασίας τοπικά και που ενισχύει αυτή η κατάσταση τη χώρα. Κατά την άποψή μου, αυτή θα είναι η προτεραιότητα, αυτή θα είναι η δική μου προτεραιότητα. Ένας από τους λόγους για τον ευάλωτο χαρακτήρα της χώρας που το εκμεταλλεύεται αυτό το γεγονός γειτονική χώρα αυτό οφείλεται στην έλλειψη ισχυρή οικονομίας και θα κάνω ό,τι μπορώ για να τους εντάξω όσο το δυνατόν στι περισσότερε ευρωπαϊκές πολιτικές, στο βαθμό του δυνατού, κυρίως όσον αφορά την ανάπτυξη υποδομών ή την προώθηση των επενδύσεων. Σχετικά με τους γεωπολιτικούς στόχους, θα πρέπει να θέλουμε να δημιουργήσουμε σταθερότητα στην ανατολική γειτονία και ασφάλεια. Επ' αυτού θα εργαστώ μαζί με τον Γιώζεφ Μπορέλ. Ευχαριστώ. Συμπληρωματική ερώτηση, Άντρος Καβίλιους. Δεύτερη ερώτηση. Συγκεκριμένα θέματα. Μολδαβία. Όπως ξέρετε, η, η κυβέρνηση ανετράπη διότι ήθελε να καταπολεμήσει η Πρωθυπουργό τη διαφθορά, να εφαρμόσει το κράτος δικαίου στη χώρα. Αυτό αναμενόταν από πολλούς στη Μολδαβία. Δυστυχώς κατέρευσε όμως ο συνασπισμό. Και έχουμε την κατάσταση που έχουμε. Και δεν έχουμε πολιτική σταθερότητα στη Μολδαβία. Αν επικυρωθεί η θέση σας, θα είναι η πρώτη κρίση που πρέπει να αντιμετωπίσετε. Πώς θα βοηθήσετε την απεμπλοκή της καταστάσεω χωρίς να υπονομεύει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και το μέλλον της Μολδαβίας για να έχετε μεγαλύτερη μόχλευση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παγώσει την οικονομική βοήθεια αν η Μολδαβία δεν εφαρμόσει σωστά τις ε, μεταρρυθμίσεις. Κύριε Βερχέη, ένα λεπτό. Ξέρω τις πρόσφατες εξελίξεις. Δεν είναι ιδιαίτερα ευτυχής για τη Μολδαβία. Θα εργαστώ συνεργαζόμενος με τη Μολδαβία για τη Μολδαβία ούτως ώστε να μην σταματήσουν οι μεταρρυθμίσεις ή να μην υπάρχει ε, πιστοχώρηση. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ακόμα και αν υπάρχει εσωτερική κρίση οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν. Εάν δεν γίνει αυτό, θα πρέπει να αναστείλουμε την οικονομική βοήθεια, όπως έγινε και στο παρελθόν. Είναι σαφές ότι η οικονομική βοήθεια συνδέεται με πρόοδο και μεταρρυθμίσεις. Και αυτό είναι κάτι μη διαπραγματεύσιμο. Ευχαριστώ. Δεύτερος ομιλητής από τους ε, σοσιαλιστές, ο κύριος Μπέντ Λάγκε, πρόεδρος ε, της ε, Επιτροπής ΙΝΤΑ, Εθνούς Εμπορίου, με την οποία έχουμε πάντοτε εξαιρετικέ σχέσεις ως Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Παρακαλώ, κύριε Λάγκε. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιο Επίτροπε, ως πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου ασχολούμαι σε βάθος με τα ζητήματα που αφορούν τη μακροοικονομική χρηματοδότηση, τις ε, συμφωνίες ε, ελευθέρων συναλλαγών και τα συναφή θέματα. Στο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των ε, δικαιωμάτων των μειονοτήτων, στο ζήτημα της ελευθερίας έκφρασης, της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος. Όλα αυτά αποτελούν ε, προτεραιότητες ε, στην, για την δική μας ατζέντα. Εσείς προέρχεστε από την διοίκηση της κυβέρνησης του κυρίου Όρμπαν που πολύ συχνά έχει υιοθετήσει θέσεις αντίθετες με τις γενικές ε, ευρωπαϊκές οπτικές. Τι εγχέγγυα κομίζεται για να μας διασφαλίσετε ότι ε, εσείς θα ακολουθήσετε στον ίδιο δρόμο των ευρωπαϊκών αξιών όπως έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Κύριε Υποψήφιο Επίτροπε, έχετε δύο λεπτά. Ως Επίτροπος, είμαι υποχρεωμένος να ακολουθώ τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σύνολο ε, συνεργασιών αλλά και προϋποθέσεων όσον αφορά την, τον σεβασμό τη ελευθερία του τύπου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη ανεξαρτησία της δικαιοσύνη. Εγώ προτίθεμαι να ε, ακολουθήσω τον ίδιο δρόμο και θα εξασφαλίσω ότι σε όλες τις σχέσεις μας θα τηρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Αυτά είναι τα συμφέροντά μας και ως Ευρωπαίος Επίτροπος ε, θα έχω υποχρέωση να υπερασπίζομαι τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια συμπληρωματική ερώτηση κύριε Λάγκη θέλετε να θέσετε. Ναι, Κύριε Βαρέλη, ε, φανταστείτε ότι υπάρχει μια υποψήφια χώρα που όπου εμφανίζονται εξελίξεις που θα μπορούσαν να υπαρθούν στο άρθρο 7. Τι μέτρα ακριβώς θα λάβετε σε μια τέτοια περίπτωση, τι ακριβώς θα κάνετε. Κύριε Βαρέλη, για, για ένα λεπτό. Στη διαδικασία διεύρυνση έχουμε την αρχή πρώτα τα θεμελιώδη. Αυτό σημαίνει ότι αν δεν σημειώνεται πρόοδος ε, στην, ε, στους αν αυτούς, ανεξαρτησία δικαιοσύνης, ανθρώπινα δικαιώματα, κράτο δικαίου, τότε μπορούν να σταματήσουν οι διαπραγματεύσει. Μπορεί ακόμη και να, να μην κλείσουν συγκεκριμένα κεφάλαια ή να ανασταλεί η να ανασταλει Εγώ δεν θέλω να ε, χρησιμοποιήσω, αλλά δεν δε θα φοβηθώ κιόλα να χρησιμοποιήσω αυτά τα εργαλεία σε περίπτωση που χρειαστεί, εφόσον δεν τηρούνται συγκεκριμένε προϋποθέσεις. Πάμε τώρα ε, στην ομάδα Renew Europe. Ευχαριστώ πολύ. Λέω ο κύριος Αστρεβίτσιος. Ε, οι εξελίξεις, ε, το εργαλείο της γειτονίας ε, σε αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και στα ανθρώπινα δικαιώματα και μεταξύ άλλων στα κριτήρια τη πυρηνική ασφάλεια. Αυτέ είναι βασικέ προποθέσει για να χορηγείται οικονομική βοήθεια σε γειτονικέ και άλλε τρίτε χώρε. Εσεί την αιρεσιμότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πώς σκοπεύετε να την εφαρμόσετε, κυρίως σε χώρες όπου παραπιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, θα ε, συμφωνήσετε να παγώσουν τα κεφάλαια, να μην δίδονται θεωρήσεις σε άτομα που ε, παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα, παραβιάζουν και την εθνική κυριαρχία των άλλων κρατών. Ο κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες, οι οποίοι έχουν συμβάλει σε Τέτοιου καταστάσεις μέσω της διαφθορά και μέσω εγκλημάτων ανά τον κόσμο. Ο κύριος ε, υποψήφιος επίτροπος, παρακαλώ για δύο λεπτά όσον αφορά το θέμα της ε, πυρηνικής ασφάλειας ε, και της ε, Λευκορωσίας. Νομίζω ότι είναι απόλυτα σαφές ότι οφείλουμε να διασφαλίζουμε την πυρηνική ασφάλεια, γιατί ακριβώς αυτός είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο στο έδαφος της, αλλά και στην γειτονιά της. Πρέπει να συνεχίσουμε τη Λευκορωσία, να διασφαλιστεί αυτή η αρχή. Η Λευκορωσία τον τελευταίο καιρό δείχνει πνεύμα συνεργασίας, έχει καταθέσει ένα εθνικό πρόγραμμα έχει συμφωνήσει να ε, γίνει μια ανάλογη έκθεση, ένα peer review, ακόμα υπολείπονται αρκετά. Οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι δικοί μας οι εμπειρογνώμονες θα πρέπει να μπορούν να μεταβούν επί τόπου να διασφαλίσουν ότι η πυρηνική ασφάλεια εξασφαλίζεται με βάση τις δικές μας αρχές. Εγώ θα δουλέψω γι' αυτό. Και όσον αφορά τις κυρώσεις για ανθρώπινα δικαιώματα, οι κυρώσεις στην εξωτερική πολιτική είναι το πιο σκληρό εργαλείο που μπορεί κανεί να εφαρμόσει. Γι' αυτό λοιπόν πριν επιβληθούν κυρώσει, ε, υπάρχουν άλλα στοιχεία ε, τα οποία μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει. Εγώ θα ήθελα ε, πρώτα απ' όλα να καταφύγω σε άλλα εργαλεία που θα έχω στη διάθεσή μου, όπως η αναστολή της χρηματοδότησης, ο διάλογος με αυτές τις χώρες. Η επιβολή των κυρώσεων πρέπει πάντα να είναι η έσχατη λύση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα και πρέπει πρώτα απ' όλα να πείσουμε τα κράτη-μέλη για να εφαρμοστεί αυτό. Εάν υπάρξει σχετική πρόταση από οποία από μία ομάδα κρατών, ευχαρίστως να το δω και εγώ για να δούμε τι είδου ωφέλη μπορεί να αποφέρει ένα τέτοιο σύστημα. Ε, συμπληρωματική ερώτηση, παρακαλώ. Ξέρουμε πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι το θέμα των κυρώσεων, αλλά η παλιά πολιτική δεν έχει αλλάξει. Εξακολουθούμε να έχουμε αυτό που λέμε ε, καρότο και ζάχαρη σχετικά με την list, ε, τον κατάλογο μαγνήσκη, αυτή τη σχετική ε, πράξη. Εσείς θα είσαστε αυστηρός στον εφαρμόζονται παντού τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα τιμωρείται άτομα και χώρες οι οποίες ε, συστηματικά παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για ένα λεπτό. Νομίζω ότι η εισαγωγή του καθεστώτος των ε, κυρώσεων είναι ένα πολύ ε, σκληρό εργαλείο και απαιτεί σύνεση, νυφαλιότητα, Προς το παρόν δεν υπάρχει τέτοια πρόταση και γι' αυτό πρέπει, αν τελικά κατατεθεί μια τέτοια πρόταση, να εξετάσουμε και όλες τις επιπτώσεις. Αυτή τη στιγμή ε, προσπαθούμε να επιτύχουμε τους στόχους μας με λιγότερο αυστηρά μέτρα και εργαλεία. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι, παραδείγματος χάνει για εγκλήματα πολέμου ήδη έχουμε τη δυνατότητα να εισάγουμε τέτοιου είδους ε, κυρώσεις. Γι' αυτό λοιπόν ίσως να μην κριθεί απαραίτητο να ληφθούν περαιτέρω κυρώσεις ε, και να μπορούμε ίσως ε, να καταφύγουμε στα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας και εκεί ίσως πράγματι να πρέπει να συμπεριληφθούν και κυρώσεις έναντι μεμονωμένων ατόμων ε, τα οποία έχουν προβεί σε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σας ευχαριστώ. ΕΛΚ. Ο κ. Βαγγέλης Μημαράκης. Για ένα λεπτό παρακαλώ, κ. Μημαράκη. Πρόεδρε, από τις εξεγέρσεις της Αραβικής Άνοιξης, οι χώρες της Νότιας Μεσογείου έχουν χαράξει διαφορετικές πορείες και κατευθύνσεις. Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξ αρχής είχε ταχθεί υπέρ των δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων με έμφαση στα ανθρώπινα δικαιώματα, αυξάνοντας μάλιστα την οικονομική της στήριξη, τώρα σχεδόν ε, εννέα χρόνια μετά η κατάσταση δεν είναι καθόλου ενθαρρυντική. Πώς αξιολογείται λοιπόν το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια και ποιες είναι οι προτεραιότητές σας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κατάστασης και πώς σκοπεύετε να διασφαλίσετε ακόμα μεγαλύτερη υποστήριξη στην περιοχή τόσο από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από τα κράτη-μέλη. Για δύο λεπτά, κύριε υποψηφία, επίτροπε. Ζητώ συγγνώμη από το αξιότιμο Ευρωβουλευτή. Την αρχή της ερωτήσεώς σας δεν κατανόησα. Για ποια περιοχή μιλήσατε. Δεν έπιασα το πρώτο κομμάτι τη ερώτησή σας. Μικρόφωνο σα παρακαλώ. Την Αραβική Άνοιξη στις χώρες της Νότιας Μεσογείου. Thank you. Σας ευχαριστώ. Είδαμε ότι η Αραβική Άνοιξη επίσης επέφερε αναταραχή στην περιοχή και βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτού. Από την άλλη πλευρά επίσης έχουμε δει ότι μπορεί να φέρει και τη δημοκρατία πιο κοντά στη γειτονιά μας, όπως στην περίπτωση της Ισίας. Θα ήθελα να συνεργαστώ με όλες τις χώρες της περιοχής και όπως είπα Παράδειγμά μου θα ήταν η Τινησία και το Μαρόκο, όπου βλέπω μεγάλη ευκαιρία, μεγάλες ευκαιρίες να συνεχιστεί και να αυξηθεί η συνεργασία μας μαζί τους και να βοηθήσουμε να παγιώσουν τις μεταρρυθμίσεις. Στον αφορά την Τινησία υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα, μεγαλύτερο δυναμικό. Είχαμε δημοκρατικές εκλογές και τώρα πρέπει να βοηθήσουμε την Τινησία να οικοδομήσει μια εύρυθμα λειτουργούσα δημόσια διοίκηση και μπορεί να χρησιμοποιεί τη χρηματοδότησή μας και που θα είναι ικανή να συνεχίσει την εφαρμογή δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και την εφαρμογή του κράτους δικαίου. Θα φροντίσω λοιπόν ούτω ώστε να παράσχουμε κάθε βοήθεια, όχι μόνο οικονομική, αλλά και τεχνογνωσία, τεχνική αρρωγή από τη στιγμή που θα υπάρχει κυβέρνηση στην Τινησία, αλλά και με τον νέο πρόεδρο της Τινησίας να τους βοηθήσω να δημιουργήσουν μια διοίκηση που θα λειτουργεί για τον λαό της Τινησίας. Συμπληρωματική ερώτηση παρακαλώ. Η κρατία, οι ελεύθερες εκλογές αποτελούν, όπως έχουμε ξαναπεί, θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες. Υπ' αυτό το πρίσμα και κάθε χρόνο πάρα πολλοί συνάδελφοι συμμετέχουν σε διάφορες αποστολές ως παρατηρητές των εκλογών ανά την Ιφίλιο. Στις χώρες της ε, Νοτίου Μεσογείου, πολλές από τις οποίες δεν έχουν παράδοση ελεύθερων και δίκαιων εκλογών, οι κυβερνήσεις αγωνίζονται να ακολουθήσουν μια δημοκρατική πορεία σύμφωνα με τις ελπίδες και τις προσδοκίες των λαών τους. Η Τινησία, όπως είπατε κι εσείς, είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα και χαίρομαι που το αναφέρατε. Η Αλγερία, στην οποία ακολουθούν προεδρικές εκλογέ το Δεκέμβριο, κάνει σημαντικές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση. Πώς κρίνετε, λοιπόν την πορεία της δημοκρατίας στις χώρες τη περιοχή και ποιες πολιτικές θα ακολουθήσετε για να ενισχύσουμε περαιτέρω τις μεταρρυθμιστικές τους προσπάθειε One minute, Commissioner Designate. Για ένα λεπτό κύριε υποψήφιε επίτροπε. Θεωρώ ότι οι αποστολές για παρατήρηση των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι εξαιρετικά χρήσιμες και θα ενεθάρρυνα όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συνεχίσουν να συμμετέχουν σε αυτές. Διότι αυτό όχι μόνο παρέχει επιτόπια γνώση για το πώς ακολουθούνται δημοκρατικοί κανόνες και γίνονται σεβαστοί καθ' όλη τη διάρκεια, αλλά δημιουργεί και πολλές ευκαιρίες Επαφή με αυτόν των χωρών σε όλα τα επίπεδα και θα ήθελα να βασιστώ στην υποστήριξή σας για τη συμμετοχή σε αυτές τι αποστολέ. και με μεγάλη χαρά σας βοηθήσω αν μπορώ με οτιδήποτε χρειαστείτε σχετικά με αυτό. Για την Αλγερία, ναι, υπάρχουν ενθαρρυντικές εξελίξεις όσον αφορά τι επικείμενε εκλογές που θα γίνουν το Δεκέμβριο. Αλλά η ιστορία της Αλγερίας μας δείχνει ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όσον αφορά τη συζήτηση των εσωτερικών υποθέσεων της Αλγερίας. Εκτός Αλγερίας θα τους ενθαρρύνουμε βεβαίως να προχωρήσουν, να ακολουθήσουν δημοκρατικό μονοπάτι, αλλά ο αλγερινός λαός πρέπει να πάει τις αποφάσεις του. Ευχαριστούμε. Από τους σοσιαλιστές, ο κύριος Ραφαέλ Τουξμάν. Ευχαριστώ κύριε υποψήφιε επίτροπε. Ο Πιέρ Ρεβερντή Γάλλος ποετής είπε δεν υπάρχει ερώτας και αγάπη, υπάρχει μόνο απόδειξη ερώτα και αγάπης. Το ίδιο ισχύει και την ανεξαρτησία. Ο συνάδελφός μου, ο Ερνέστο Ορτασούν, ε, ζήτησε απόδειξη ανεξαρτησίας. Όχι ομιλία για ανεξαρτησία, απόδειξη ανεξαρτησίας. Μιλάει για τη θέση σας ο κ. Ορμπάν εάν αποδείξετε ότι είσαι ανεξάρτητος θα σα υποστηρίζαμε. Επαναλαμβάνω το ίδιο ερώτημα. Χρειαζόμαστε απόδειξη ανεξαρτησίας. Καταδικάστε τη φράση που είπε ο κύριος Ορμπάν. Μπορείτε να καταδικάσετε επίσης και την έννοια της μη φιλελεύθερης δημοκρατίας που αναφέρθηκε στην Ουγγαρία, που είναι το αντίθετο των αρχών που πρέπει να προωθούμε στην πολιτική της γειτονίας. Κύριε υποψήφιε επίτροπε, για δύο λεπτά. Απόδειξη της ανεξαρτησίας μου είναι το έργο που έχω επιτελέσει ε, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για τέσσερα χρόνια ήμουνα επικεφαλής μονάδας που είχε ως καθήκον, ένα καθήκον μάλλον το οποίο ήταν αδύνατον να επιτευχθεί για 40 χρόνια και συνέβαλα στο να στεφτεί με επιτυχία η διαδικασία αυτή. Παρά τι πολύ βαριές και πολύ δύσκολες διαπραγματεύσει που χρειάστηκε να γίνουν με πολλά κράτη-μέλη. Κατάφερα και χειρίστηκα το ζήτημα αυτό με ανεξάρτητο τρόπο, χωρίς καμία εξωτερική παρέμβαση. Αυτό για μένα αποτελεί απόδειξη απτή των ικανοτήτων μου να ενεργώ και να, δράτω, και να πράττω με ανεξαρτησία. Όσον αφορά τις δηλώσεις κυβερνήσεων, αυτές είναι ευθύνη των ίδιων των κυβερνήσεων. Εγώ ως Επίτροπος θα τηρώ τη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε πνεύμα συναδελφικότητας και συνεργασίας με τους ε, συναδέλφους μου στο Σώμα των Επιτρόπων. <coughs> ερώτηση, κύριε Γκλούξμαν. Δεν θέλετε να καταδικάσετε συγκεκριμένη φράση που είπε ο κ. ούτε την έννοια της μη φιλελεύθερης δημοκρατίας να πω κάτι. Ένας μεθανάστη δημιουργεί τρομοκρατική απειλή για την ασφάλεια τη δημοκρατική, είπε ο κ. Ορμπάν. Ερώτηση. Εφόσον η Ουγγαρία καταδικάστηκε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε στην Ουγγαρία στο δικαστήριο για δίδυση μορφών την δημοσιοσία το δικαίωμα ασύλου και επιστροφής όσον αφορά το δίκαιο της Ένωσης. Τι θα κάνετε για να ασκηθεί μια πολιτική στην πολιτική γειτονίας και που εφαρμόζει η Ουγγαρία αντίθετη από αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ε, όσον αφορά το άσυλο και τη μετανάστευση. Υπάρχει αντίθεση μεταξύ της κυβερνήσεώς σας και της πολιτικής της Ευρωπαϊκής. Τι θα κάνετε γι' αυτό. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό κύριε υποψήφιο επίτροπε. Το χαρτοφυλάκιο μου θα ε, περιλαμβάνει και θα καλύπτει τις ε, ε εξωτερικές διαστάσεις του χαρτοφυλακίου της μετανάστευσης. Εκεί θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι τη γραμμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ότι πρέπει να βοηθήσουμε τις, ε, τους γείτονές μας στη, στην Ανατολή και στον Νότο να προστατεύσουν τα εξωτερικά τους σύνορα, να ε, αντιμετωπίσουν την παράνομη μετανάστευση, αλλά να ε, ταυτόχρονα φροντίσουν και τους μετανάστες που βρίσκονται στην επικράτειά τους. Και ε, εγώ θα συνεχίσω, όπως και η προηγούμενη Κομισιόν, να επιτελώ αυτό το ε, καθήκον. Αυτή είναι η πολιτική που εκπροσωπώ εγώ, αυτή είναι η πολιτική που θα ακολουθήσω στη διάρκεια της θητείας μου. Ευχαριστώ. Εκ μέρους των Πρασίνων. Εκ μέρους ε, των Πρασίνων κυβέρνησή σας ήταν εξαιρετικά φιλική προς τον κύριο Πούτιν. Τέσσερις επισκέψεις έχουν γίνει. Η Ουγγρική κυβέρνηση ε, επέτρεψε μάλιστα στην Ρωσική Τράπεζα Επενδύσεων να δραστηριοποιηθεί στην Ουγγαρία με πλήρη ασυλία. Τα, το, τα μέλη του προσωπικού αυτής της τράπεζας έχουν διπλωματικά διαβατήρια και δεν ελέγχονται από τις διαδικασίες του, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς θα μπορέσετε εσείς να αντιταχθείτε στη ρωσική επιρροή στην περιοχή της Ανατολικής Γειτονίας και στα Δυτικά Βαλκάνια όταν η δική σας κυβέρνηση ενεργά προώθησε και ε, υποστήριξε τα ρωσικά συμφέροντα εντός της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά κύριε υποψήφια επίτροπε έχετε. Ευχαριστώ. Καθήκον ενός ε, επιτρόπου ε, δεν είναι να υπερασπιστεί μια συγκεκριμένη εθνική γραμμή και δεν θα το πράξω εγώ. Ούτε της Ουγγαρίας, ούτε καμίας άλλης χώρας. Καθήκον μου θα είναι να προασπίσω την ευρωπαϊκή πολιτική την οποία συνδιαμορφώνει το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Αυτή θα είναι η δουλειά μου. Όπως είπα και νωρίτερα, το έχω κάνει αυτό για τέσσερα χρόνια. Μου ανατέθηκε ε, από την Κομισιόν να αναλάβω ένα πολύ ευαίσθητο φάκελο, να υπησέλθω σε πολύ ευαίσθητες και λεπτές πολιτικές συζητήσεις και τις ε, ολοκλήρωσα με επιτυχία. Και αυτό μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα το πράξω και αν μου αναθέσετε το, τη θέση του Επιτρόπου. Συμπληρωματική ερώτηση. Το Κρεμλίνο υποστηρίζει προπαγάνδα και στο διαδίκτυο και στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης, επηρεάζοντας τα κράτη-μέλη αλλά και τη γειτονία μας. Αυτή η εκστρατεία παραπληροφόρησης είχαν καταστροφικές, είχε καταστροφικές απο, καταστροφικά αποτελέσματα για τη δημοκρατία. Αν εσείς επιβεβαιωθείτε ως επίτροπος, πώς θα στηρίξετε Γεωργία, Μολδαβία, Ουκρανία για να καταπολεμήσουν ε, ε, την υβριδική αυτή απειλή. Ακόμα και στην Ουγγαρία, κρατικά μέσα ενημέρωσης διασπείρουν ψευδείς ειδήσει οι οποίες προέρχονται από την ε, Ρωσία. Πώς το σχολιάζετε αυτό. Κύριε Βαρχέη, εγώ θα συνεργαστώ με τον Γιώζε Μπορέλ στον τομέα αυτό έχουμε δημιουργήσει στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης την ε, στρατηγική ομάδα επικοινωνίας, η οποία ήδη έχει ορισμένες επιτυχίες όσον αφορά την απόκρουση των υβριδικών απειλών και των ψευδών ειδήσεων. Και θα συνεργαστώ με τον ύπατο εκπρόσωπο, ε, ιδίως στην ε, Ουκρανία, γιατί εκεί διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο όπου επηρεάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και η κοινή γνώμη. Και θα αξιοποιήσω όλα τα χρηματοδοτικά μέσα που θα έχουμε στη διάθεσή μας, ώστε η Ουκρανία να μπορέσει να καταπολεμήσει το φαινόμενο αυτό. Thank you. Πολύ ωραία ε, για την ομάδα ID Jérôme Rivier. Κύριε υποψήφιε επίτροπε, επαναλαμβάνουμε βέβαια κάποια πράγματα, δύο θέματα που με αφορούν και με ενδιαφέρουν τα Δυτικά Βαλκάνια και η Τουρκία. Αναφερθήκατε στις παράνομες γεωτρήσεις στα κυπριακά χωρικά ύδατα των Τούρκων και τα προβλήματα στη Συρία και την εισβολή. Και έχουμε βέβαια και την κατοχή της, το 1974 Κύπρου και, και έχουν ανακήρυξει ε, επίσης μια δημοκρατία που αναγνωρίζει το κάνει στη, στη Βόρεια Κύπρο και η πολιτική του Ερντογάν δημοσ... Ε, είχε, χρησιμοποιούσε έσοδα από το πετρέλαιο και χρησιμοποιούσε την Ισλαμιστική τρομοκρατία σε όλη την Ευρώπη. Συζητούσαμε στο Μικύκλιο αυτές τις παράνομες γεωτρήσεις και από όλε τι ομάδε είχαμε ομοφωνία, θέλαμε να καταγγείλουμε την Τουρκία γι' αυτό και να καταδικάσουμε. Το ερώτημα είναι πώ θα θέσουμε τέρμα σε αυτή την πολιτική που είναι η πολιτική σαδομαζοχιστική που επικρατεί ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρκία. Η Τουρκία απειλεί, επιτίθεται και εμεί πληρώνουμε και πληρώνουμε ακόμα. Δεν ήρθε η ώρα να σταματήσουμε με αυτό το, το ψέμα τη ενδεχόμενη προσχώρηση και να μην ε, σπαταλάμε πλέον τα δισεκατομμύρια που του στέλνουμε. Ο κύριος υποψήφιος ε, για δύο λεπτά. Όσον αφορά στη διαδικασία ένταξης της Τουρκίας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, βλέπουμε ότι ήδη υπάρχει στασιμότητα. Βέβαια, το να πάψουν οι διαπραγματεύσεις ε, χωρίς να υπάρξει ένταξη, αυτή είναι μια πολύ σημαντική στρατηγική απόφαση που θα ληφθεί από το Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αποφασίσει ένας ε, επίτροπος. Ως εκ τούτου θα υπάρξει ουσιαστική συζήτηση για τις μελλοντικές μας σχέσεις με την Τουρκία και βεβαίως αυτό θα είναι ένα στρατηγικό ερώτημα που θα πρέπει να εξετάσουμε. Από την άλλη βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Τουρκία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σύμμαχος ε, του ΝΑΤΟ και έχει 100 εκατομμύρια περίπου κατοίκους, μια πολύ μεγάλη χώρα και κατ' ουσίαν ε, στη δική μας τη γειτονιά. Άρα δηλαδή όταν αξιολογούμε τις ε, μελλοντικές μας σχέσεις, οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη μας όλους τους ε, παράγοντες. Ένας από αυτών των παραγόντων είναι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Συμπληρωματική ερώτηση παρακαλώ. Ε, σας ευχαριστώ όσον αφορά τα Βαλκάνια και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τη διεύρυνση, φαίνεται περίπου συνέχεια να φουσκώνουμε ένα μπαλόνι, με αυτό μοιάζει. Και το συνέστημά μας είναι ότι αυτό τελικά θα εκραγεί. Ο πρόεδρος Μακρόν υπό την πίεση της κυρίας Λεπέν ανήκουσε, με, ε, ε, ε, εκπροσωπούν πολλούς, πολλά εκατομμύρια πολιτών που δεν θέλουν πλέον αυτή την πολιτική και είναι αντίθετη να μπει η Βόρεια Μακεδονία και η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Με αντικείμενου λόγου ε, ε, ε, υπάρχει πολιτική, είναι εύθραστη ε, χώρε, έχουμε προβλήματα στο κοσμοπέδιο και η Σερβία έχει ιστορική ιστορία που δεν δείχνει ότι έχει δυτική λογική. Θέλετε να τονίσετε, είπατε, τη μεταρρύθμιση, τι αναγκαίε μεταρρυθμίσει αυτές αυτέ τι χώρε. Μπορείτε να αντισταθείτε στην πλειοψηφία τη πλειοψηφία εδώ που πανικοβάλλεται και κινείται κατά των λαών σε μια φρενήρη α, κούρσα προ μεγαλύτερη διεύρυνση. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ. Για ένα λεπτό παρακαλώ. Το δικό μου το καθήκον ως Επίτροπος ε, Αρμόδιος για τη διεύρυνση θα είναι όχι μόνο να πείσω τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων για τις δικές μας τις ε, προϋποθέσεις και να συμμορφωθούν με αυτές, αλλά να πείσω και τα κράτη-μέλη και τους πολίτες μας ότι ε, όλα αυτά είναι προς το δικό μας συμφέρον, κυρίως ε, το να εκπληρώνονται ε, το να τηρούνται οι κανόνες, να εκπληρούνται οι προϋποθέσεις. Άρα δηλαδή η γέφυρα ανάμεσα στα κράτη-μέλη και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Και να είστε σίγουρος ότι ε, θα υπερασπιστώ τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην περιοχή με σθένος, έτσι ώστε να εξεταστούν όλες οι πτυχές των προβλημάτων, αλλά θα τους προσφέρουμε και κίνητρα, έτσι ώστε οι χώρες αυτές να αναπτυχθούν περαιτέρω και να έρθουν πιο κοντά μας και αυτό είναι ένα τμήμα της πολιτικής που επιτιμώ να εφαρμόσω. Και νομίζω με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη μας όλες τις υφιστάμενες ανησυχίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ο κύριο Τζαμπάτσκι εκ μέρους του ε, ECR, αλλά δεν τον βλέπω, δεν είναι παρόν στην αίθουσα. Μήπως θέλει ανταυτού να λάβει κάποιος άλλος το λόγο εκ μέρους του ECR. Νάτος, εδώ είναι κύριε Τζαμπάτσκι. Μήπως ε, μπορείτε να μας πείτε το όνομά σας, αλλά βεβαίως έχετε το λόγο. Θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα στα Ολλανδικά. Λοιπόν, για τη Μεσόγειο και το Λίβανο μιλήσατε και για άλλε χώρες. Δεν άκουσα πολλά όμω όταν μιλήσατε για χώρες δεν αναφερθήκατε στο Ισραήλ. Μπορείτε να μας πείτε κάποια πράγματα για το Ισραήλ. Ποια είναι η άποψή σας για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκή Ενώσεω και Ισραήλ. Πώς μπορούν να ενισχυθούν οι σχέσεις κατά την άποψή σας. Έχουμε συμφωνία σύνδεση με το Ισραήλ και χρειάστηκαν πολλά χρόνια διαπραγμάτευσης. Θα ήθελα να μου πείτε τι πιστεύετε για τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ. Σας ευχαριστώ. Για δύο λεπτά κύριε υποψήφια επιτρόπε. Ευχαριστώ πολύ. Πράγματι έχουμε συμφωνία σύνδεσης με το Ισραήλ. Έξοχες εμπορικές σχέσεις έχουμε με το Ισραήλ και πολύ υψηλό επίπεδο συνεργασίας σε πάμπολους τομείς όπως Φερρυπίν έρευνα και ανάπτυξη. Αυτό είναι σημαντικότατο. Πρέπει να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε το επίπεδο συνεργασίας σε όλους αυτούς τους τομείς. Όμως, έχουμε επίσης και κάποια προβλήματα σε σχέσει μα όσον αφορά τη ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή και τη σχέση του Ισραήλ με την Παλαιστίνη και τι κα... κατεχόμενε περιοχέ. Εκεί ξεκολουθώ να υπερασπίζουμε τη γραμμή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, ότι μόνο μια λύση δύο κρατών μπορεί να δώσει μακροχρόνια ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε συνεργαζόμενοι με το Ισραήλ και την Παλαιστίνη να το πετύχουμε αυτό. Βέβαια αυτό δεν είναι πρωταρχικά δική μου ευθύνη, αλλά πρωταρχική ευθύνη του Ζωζεφ Μπορέλ, διότι στο κάτω-κάτω είναι σημαντικό θέμα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας. Όμως έχω εργαλεία στη διάθεσή μου ούτω ώστε να ενθαρρύνω την ε, διαδικασία, αλλά και να σταθώ στο πλευρό των Παλαιστινιακών αρχών και να ξεκολουθώ να βοηθώ το έργο τους όσον αφορά το θέμα των προσφύγων ή ε, την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας που παρέχουμε. Δυστυχώς είδαμε και ατυχείς εξελίξεις πρόσφατα σε σχέση με έναν από τους, τους βασικούς οργανισμούς στην περιοχή. Ελπίζουμε να διευθωθεί η κατάσταση το ταχύτερο δυνατόν στο UNRWA και θα καθίσουμε συνεργαζόμενοι μαζί τους και θα συνεχίσουμε τη χρηματοδότηση αυτής της οργανώσεως μόνο από τη στιγμή που όλες οι ατασταλείς και τα προβλήματα θα ρυθμιστούν απόλυτα. Πρέπει να συνεχίσουμε τις επαφές με αυτούς, διότι είναι βασικός φορέας επιτόπιος. Ε, για ένα λεπτό έχετε το χρόνο τώρα για μια συμπληρωματική ερώτηση. Ε, eh, eh, Ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας και τις ε, δοθήσεις εξηγήσεις. Μια συμπληρωματική ερώτηση αν επιτρέπετε. Συμφωνείτε μαζί μου ότι το Ισραήλ είναι απειλούμενο λόγω πιέσεων που ασκούνται από το Ιράν. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτό το θέμα, ποιος έχει ευθύνη, μήπως θα ήταν δυνατό στα πλαίσια του χαρτοφυλακίου σας να δείτε πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε την, τα προβλήματα ασφαλείας που ε, αντιμετωπίζει το Ισραήλ και τις απειλές που αντιμετωπίζει το Ισραήλ. Ε, νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα μπορούσατε να το εξετάσετε. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, ένα λεπτό για να απαντήσετε. Η γραμμή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως πάντα ήταν η εξή ότι δεν δεχόμαστε καμία απειλή εναντίον της ασφαλείας του Ισραήλ. Εάν επικυρωθεί θέση μου, διορισμός μου σαν επίτροπος, αυτή τη γραμμή θα πρέπει να επιδιώξουμε. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η αδίποτη εξωτερική απειλή και εσωτερική, είτε από τα κατεχόμενα είτε από έξω από το Ισραήλ, δεν θα πρέπει μόνο να καταδικάζονται αυτές οι απειλές, αλλά να απορρίπτονται όσον αφορά τη σχέση με το Ιράν, δεν εμπίπτει στο χαρτοφυλάκιό μου Άρα δεν θα ήταν σωστό να σας δώσω συγκεκριμένη απάντηση από αυτού. Αυτό που είμαι έτοιμος να κάνω είναι όπως προανέφερα. Είμαι έτοιμος να παράσχω κάθε αναγκαία βοήθεια που εντάσσεται στο χαρτοφυλάκιό μου, ώστε να εγγυηθώ την ασφάλεια του Ισραήλ. Thank you for the EPP. Ευχαριστώ για το ΕΛΚ, ο κύριος Λουκάς Μάντελ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, το ερώτημά μου αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια και την ε, φυγή εγκεφάλων από τα Δυτικά Βαλκάνια. Καταρχάς βεβαίως θα ήθελα να σας συγχαρώ για τον ε, ορισμό σας, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι πάντοτε τιμή να έχει κανείς την ε, ευκαιρία να υπηρετήσει τους Ευρωπαίους πολίτες από μια τέτοια θέση. Δεύτερον, χαίρομαι που με σαφήνεια ε, τονίσατε την κριτική που ασκήσατε στην ε, ε, τουρκική εισβολή στη Συρία και που υπογραμμίσατε τις ανησυχίες που πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει απέναντι στη στάση της Τουρκίας λόγω των αρνητικών εξελίξεων των τελευταίων εβδομάδων. Και αυτό συνδέεται και με έναν τρόπο με την φυγή εγκεφάλων, διότι άνθρωποι που έχουν εκπαίδευση, που έχουν μορφωτικό ε, επίπεδο υψηλό εγκαταλείπουν τα Δυτικά Βαλκάνια με προορισμό την Τουρκία, για παράδειγμα από το Κόσοβο, το οποίο εξακολουθεί να μην έχει ε, τη δυνατότητα να, οι πολίτες του να έρχονται χωρίς θεωρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει όμως μια τέτοια δυνατότητα ώστε οι άνθρωποι αυτοί να πηγαίνουν στην Τουρκία. Τι θα κάνετε εσείς ώστε να βοηθήσει τα Δυτικά Βαλκάνια να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της φυγής εγκεφάλων, του brain drain. best tool το καλύτερο εργαλείο για να αντιμετωπίσει κανείς την φυγή εγκεφάλων είναι να αναπτυχθεί η τοπική οικονομία. Μια τοπική οικονομία η οποία θα μπορεί να απασχολεί τους νέους επαγγελματίε από τις χώρες αυτές. Αλλά για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζονται πολλά πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Βασικές υποδομές, οικονομική ανάπτυξη, άμεσες ξένες επενδύσεις, ανταγωνιστικό εκπαιδευτικό σύστημα. Γι' αυτό το λόγο η Κομισιόν ήδη έχει ξεκινήσει προσπάθειες προώθησης και χρηματοδότησης της ανώτατης εκπαίδευσης και από και της επαγγελματικής κατάρτισης στην περιοχή αυτή. Τα στοιχεία βεβαίως είναι πραγματικά πολύ κρίσιμα. Κατά μέσο όρο βλέπουμε ότι 40% του πληθυσμού των Δυτικών Βαλκανίων έχει εγκαταλείψει τις ε, χώρες αυτές. Και πρόκειται βεβαίως για τους νέους ανθρώπους, για τους επαγγελματίες εκείνους πάνω στους οποίους θα μπορούσε να βασιστεί η οικονομική ανάπτυξη. Πρέπει να επαναπροσελκυστούν οι άνθρωποι αυτοί. Όμως αυτό μπορεί να γίνει μόνο εφόσον τα επόμενα πέντε χρόνια υπάρξει οικονομική ανάπτυξη στις χώρες αυτές. Βεβαίως αυτό μπορεί να γίνει ε, εις βάρος των θεμελιωδών δικαιωμάτων του κράτους δικαίου, οποιασδήποτε Βασική μα αρχή και αξία. Αυτά θα πρέπει να συμβαδίζουν. Διαφορετικά, καμία εταιρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα έχει την προθυμία να κάνει επενδύσεις και να διακινδυνεύσει τα κεφάλαιά της σε μια περιοχή η οποία είναι απρόβλεπτη. Για το καθεστώς ε, απαλλαγή από τι θεωρίες για το Κόσοβο. Δυστυχώ, η υπόθεση αυτή έχει μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο και έχει μπλοκαριστεί και στον διάλογο μεταξύ Πρίστινας και Βελιγραδίου. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε μπροστά μας μια ιστορική ευκαιρία να καταλήξουμε σε μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των δύο πρωτευουσών, ελπίζουμε ακόμη και φέτος. Αν γίνει κάτι τέτοιο, το ζήτημα της απαλλαγής των πολιτών του Κωσόβου από τις θεωρήσεις θα ξανανοίξει με νέα ορμή. Ταυτόχρονα θα πρέπει βεβαίως, συμφωνώ μαζί σας, να διευκολύνουμε την ε, δυνατότητα των ε, πολιτών του Κωσόβου να πραγματοποιούν ταξίδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Συμπληρωματική ερώτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Φιλόδοξο ε, που μας είπατε ότι μπορεί μέχρι και φέτος να επιτευχθεί μια τέτοια συμφωνία. Φαντάζομαι ότι το έχετε συνεννοηθεί αυτό και με τον κύριο Γιώζε Πορέλ. Είπατε άλλωστε ότι θέλετε να λειτουργήσετε ω γέφυρα μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Θέλετε λοιπόν να πείσετε και την ε, γαλλική κυβέρνηση για ε, μια τέτοια προοπτική για την διευκόλυνση των Δυτικών Βαλκανίων όσον αφορά τη δυνατότητα των πολιτών των χωρών αυτών να κάνουν ε, ταξίδια προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλετε, έχετε σκοπό να δημιουργήσετε και μια ομάδα επιτρόπων η οποία θα ασχολείται συγκεκριμένα και εξειδικευμένα με το ζήτημα αυτό των θεωρήσεων για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ο υποψήφιος επίτροπος. Πολύ σύντομα. Αυτά που έχω δει εγώ στο Συμβούλιο. Εγώ ήμουν παρόν στις συζητήσεις που έγιναν και φέτος και πέρσι. Πρόκειται για μια αποτυχία λόγω διαφορετικών εκτιμήσεων της ίδιας κατάστασης. Δική μου προτεραιότητα λοιπόν θα είναι να καταλήξουμε σε μια κοινή εκτίμηση και από πλευράς κρατών μελών και από πλευράς κομισιών όσον αφορά τα πραγματικά γεγονότα. Θέλω να εντάξω τα κράτη-μέλη στις ε, ερευνητικές ε, αποστολές που πραγματοποιούμε σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων ώστε να καλυφθεί ολόκληρη η περιοχή, να δούμε τα πραγματικά γεγονότα, τι εξελίξει και να καταλήξουμε σε μια κοινή εκτίμηση και αξιολόγηση, ώστε να μην υπάρξει άλλη αποτυχία. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε έναν ξεκάθαρο κατάλογο ε, στόχων που έχουν επιτευχθεί και στις δύο πλευρές, και για τα Δυτικά Βαλκάνια και για εμάς. Και έτσι δεν θα υπάρχουν εκπλήξεις στο μέλλον. Όσον αφορά το άλλο θέμα που θίξατε, που σχετίζεται με τη γαλλική κυβέρνηση, δεν είναι μόνο η γαλλική κυβέρνηση, πρέπει να σας πω. Είναι και η Ολλανδική κυβέρνηση αυτή που πρέπει να πείσω και η κυβέρνηση της Δανίας που πρέπει επίσης να πιστεί. Αλλά με χαρά θα το κάνω και από την αρχή της ανάλυσης των καθηκόντων μου θα επιδιώξω ε, μια τέτοια εξέλιξη γιατί χωρίς αυτές τις κυβερνήσεις δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε το στόχο. Εκ μέρους του Renew, Κλέμεν Γκρόσεου, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ε, κύριε υποψήφιε Επίτροπε. Η υποψήφια Πρόεδρος είπε ότι θα είναι ε, μία επιτροπή η οποία θα δίνει σημασία σε γεωπολιτικά θέματα. Εσείς πιστεύετε ότι ε, θα συνεχιστεί, ότι είναι αυτό θα παίξει σημαντικό ρόλο ή θα υπάρξουν και άλλες αξίες που θα παίξουν ρόλο στην πολιτική σας ε, στη διεύθυνση. Δηλαδή πώς ακριβώς ε, θα εξισορροπήσετε αυτές τις δύο μερικές φορές αντιμαχόμενες και αντιφατικές αρχές. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω ότι πρόκειται για αντιφατικές ε, αρχές και αντιμαχόμενες μπορούμε να έχουμε και διεύρυνση και θεμελιώδης ελευθερίες και κράτος δικαίου ε, στα Δυτικά Βαλκάνια. Γιατί χωρίς αυτά δεν μπορεί να υπάρξει διεύρυνση. Αυτό όλοι μας το γνωρίζουμε και εγώ θα συνεργαστώ στενά με τις χώρες των ε, Δυτικών Βαλκανίων αλλά και με τα δικά μας τα κρατημέλη για να γίνουν όλα αυτά πραγματικότητα. Και θα ήθελα να κατανοήσουν οι ε, χώρες ένταξης ότι αυτή είναι μια ευρεία έννοια, ε, αλλά είναι και κάτι το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο για την καθημερινή ζωή, δηλαδή για την οικονομία, για την κοινωνική ζωή, διότι αλλιώς ε, οι χώρες αυτές δεν μπορούν να έχουν μια ουσιαστική σχέση με εμά. Και χωρίς αυτό δεν μπορεί να υπάρχει εμπιστοσύνη. Άρα δηλαδή θα τις, έτσι μόνο μπορούμε να τις καλωσορίσουμε στη δική μας την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα πρέπει να εργαστούμε παράλληλα για να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες έτσι ώστε αυτές να συμμετέχουν σε περισσότερες δικές μας πολιτικές. Από την άλλη όμως να διασφαλίσουμε ότι και εκείνε δεν πρέπει να ξεχνάνε τα βασικά. Είναι σαφές από αυτά που είδαμε τον Οκτώβρη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι αν δεν τα επιδιώξουμε όλα αυτά δεν υπάρχει άλλη λύση αλλά και πάλι η ευρωπαϊκή προοπτική υπάρχει, δεν έχει αλλάξει, ε, μπορεί όμως να γίνει πραγματικότητα μόνο εφόσον καλύπτονται όλες αυτές οι προϋποθέσεις. Συμπληρωματική ερώτηση παρακαλώ. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας για το προενταξιακό εργαλείο. Ε, μεταξύ άλλων ε, χρησιμοποιήθηκε και για να αντιμετωπιστεί η μεταναστευτική κρίση. Ε, θα κάνετε κάποια αλλαγή έτσι ώστε ε, αυτό το προενταξιακό εργαλείο να βοηθήσει τις επιλέξιμες χώρες, ενώ για τη μεταναστευτική πολιτική θα εξευρεθούν άλλα πιο κατάλληλα εργαλεία. με, τις νέες, με τις νέες προτάσεις για το νέο πουδουπού είναι σαφές ότι το, η προενταξιακή βοήθεια θα χρησιμοποιείται μόνο για να στηριχθούν οι χώρες για την προετοιμασία τους για το κράτος δικαίου και για όλους τους άλλους τομείς που είναι καθοριστικοί και πρέπει να εξελιχθούν σε αυτές τις προενταξιακές χώρες. Ε, θα έχουμε και ένα άλλο εργαλείο, τις συμφωνίες ε, των ελεύθερων εμπορικών ανταλλαγών, έτσι ώστε ε, να μην μπερδεύονται αυτά τα δύο, αν βέβαια εγκριθεί το δεύτερο δεν θα υπάρχει καμία ανάμειξη ανάμεσα στο προενταξιακό, στην προενταξική βοήθεια και σε μεταναστευτικές δράσεις. Σας ευχαριστώ για τους μη εγγεγραμμένους συναδέλφους. Μάρτιν Ζεγκέση. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Συγχαίρω τον κύριο Βερχέη που τα κατάφερε μέχρι εδώ επελέγεται από μια κυβέρνηση, από ένα κόμμα που ο Κίο δρούσε επί 9 χρόνια κατά του κράτους δικαίου. Γι' αυτό έχουμε και μια διαδικασία του άρθρου 7 που έχει κινηθεί κατά της Ουγγαρίας και μπορεί να έχει σοβαρότητες συνέπειες. Διότι το Φίντες δημιουργεί ένα ε, κόμμα και ένα πολιτικό σύστημα που δυσδεί στην πολιτική διοίκηση, στη δημόσια διοίκηση, το Υπουργείο Εξωτερικών δεν εξαιρείται. Είστε γνωστός σαν στρατιώτης του Φίντες εδώ στις Βρυξέλλες παρόλο που είσαστε ένας εμπειρογνώμονα καλά προετοιμασμένος. Τι εγγύσει μας δίνετε ότι θα κινηθείτε ανεξάρτητα από το Φίντες και τον κύριο Ορμπάν, τι εγγύσει μπορείτε να μας δώσετε ότι θα εξυπηρετείτε, θα υπηρετείτε μάλλον τα συμφέροντα των Ευρωπαίων ε, πολιτών και όχι των ολιγαρχών του Φίντες. Πώς μπορείτε να συνομιλείτε με προενταξιακές χώρες και να τους ζητάτε να σέβονται κάποιες αρχές, παραδείγματος χάρη όταν η κυβέρνησή σας κινείται κατά αυτών των αρχών που υποστηρίζετε έναντι των υποψηφίων χωρών. Ευχαριστώ κύριε υποψήφιε επίτροπε. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας αγαπητέ συνάδελφε. Σύμφωνα με τις ιδρυτικές συνθήκες, κάθε μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διορίζεται από κυβερνήσει των κρατών μελών σε συμφωνία με την εκλεγήσα πρόεδρο. Αυτό ισχύει και στη δική μου περίπτωση. Δεν είμαι μέλος κανενός πολιτικού κόμματος. Πώς μπορείτε να με θεωρείτε λοιπόν σαν ε, ως κόμματος. Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση Νίκολα Γκρουεύσκη, το μόνο που μπορώ να πω είναι αυτό που είπε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και αυτό θα τηρήσω και στο μέλλον. Όπως υποσχέθηκα επανειλημμένα εδώ, σήμερα, θα δρώ εντελώς ανεξάρτητα, δεν θα λαμβάνω οδηγίες από κανένα κράτος μέλος, όπως ήδη έκανα όταν υπηρετούσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θα λάβω οδηγίες από καμία κυβέρνηση και κανένα θεσμικό όργανο θα κινούμε συλλογικά, κολεγιακά, σαν μέλος του κολεγίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη συγκεκριμένη υπόθεση που αναφέρατε τα κράτη-μέλη αποφασίζουν σχετικά με αυτό επίσης επί των κανόνων για το άσυλο και πρέπει να εφαρμόσει τους κανόνες η Ουγγαρία. Γι' αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών και δεν έχω περαιτέρω σχόλια. Ευχαριστώ. Συμπληρωματική ερώτηση, κύριε Κονσέσκη. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ για την απάντηση, κύριε Υποψήφια Επίτροπε. Σε αυτή την ε, ακρόαση αμφισβητήθηκε η ανεξαρτησία σας ή αναφέρθηκε επανειλημμένα. Και η δήλωση του κυρίου Ορμπάν στον Πακού, στο Συμβούλιο ε, αναφέρθηκε, να, δοκιμάσουμε ξανά, στον Πακού, στο Συμβούλιο με την Τουρκία, είπε και ο Σορμπάν ότι η Ουγγαρία πολεμάει για αυτό το σημαντικό χαρτοφυλάκιο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο μετά θα χρησιμοποιήσει η Ουγγαρία για να βοηθήσει τους φίλους της χώρας που είναι το Αζερβαϊτζάν και η Τουρκία. Και να προσπαθήσει να προωθήσει τα συμφέροντα των εν λόγω χωρών. Ό,τι και αν σκέφτεστε μεταξύ, το σχέση μεταξύ Αζερβαϊτζάν, Ευρωπαϊκής Ενώσης και Τουρκίας ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, σίγουρα δημιουργεί ανησυχίες αυτό ότι ένας Ευρωπαίος Επίτροπος θα χρησιμοποιηθεί από τον Πρωθυπουργό από ένα κάτω μέλο σαν μαριονέτα. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Πώς μπορείτε να μας εγγυηθείτε ότι δεν θα λάβετε οδηγίες από τον κύριο Ορμπάν. Σημαντική απάντηση κύριε Βερέη για ένα λεπτό. Κύριε Τζέγκεση, μπορώ μόνο να επαναλάβω αυτά που είπα. Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μπορούν να λαμβάνουν οδηγίες από καμία κυβέρνηση κράτους μέλους ή οποιοδήποτε άλλο θεσμό θα συμμορφωθώ με αυτό τον κανόνα, δεν θα λάβω οδηγίες και μπορώ να ακολουθώ μόνο τους κανόνες των ιδρυτικών συνθήκων, οι, οποίες, οι οποίοι κανόνες θα με κατευθύνουν και θα με προσανατολίζουν στην εργασία μου. Σαν επικεφαλής μονάδας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέδειξα τη δυνατότητα που έχω να εργάζομαι ανεξάρτητα, ανεξάρτητος από η αδίποτε εξωτερική επιρροή. Ευχαριστούμε. Επόμενο ερώτημα από τον κύριο Σίντε εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, θέλω να επανέλθω στο ζήτημα που αναφέρθηκε νωρίτερα για την αντιπροσωπεία στη Βόρεια, ε, Μακεδονία. Ως ε, εκπρόσωπος της Ουγγαρίας στο Συμβούλιο, η Ουγγαρία έδωσε άσυλο στον κύριο Νίκολα Γκρούευσκι, τον καταδικαστέντα πρώην Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας. Η Ουγγαρία δε βοήθησε στην καταδίκη, ε, στην, στην ε, φυγή καταδικαστέντος από την Ευρωπαϊκή Ένωση με διπλωματικά αυτοκίνητα. Νομίζω ότι αυτά τα ζητήματα πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διελευκαθούν πλήρως από εσάς, ιδίως όταν μιλάμε για το κράτος δικαίου. Γι' αυτό νομίζω ότι πολιτικά και νομικά είναι ασύμβατο αν δέχεστε αυτά που συνέβησαν με ευθύνη της Ουγγρικής κυβέρνηση. θέλω να μας πείτε την δική σας γνώμη για αυτήν την υπόθεση. Κύριε Βαρχέ, έχετε δύο λεπτά στη διάθεσή σας. Στην περίπτωση αυτή, όπως εξήγησα και στον Ούγγρο συμπατριώτη μου, η απόφαση χορήγησης ασύλου υπό το Ευρωπαϊκό Δίκαιο εναπόκειται ε, στα κράτη-μέλη. Ως ε, Επίτροπος, εγώ δεν θα είμαι υπεύθυνος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του χαρτοφυλλοκίου μου. Ωστόσο, δεν θα επιτρέψω σε καμία δραστηριότητα που εντάσσεται στο δικό μου χαρτοφυλάκιο να και καμία υπηρεσία να δεχτεί πράξη θεσμικού οργάνου ή κράτους μέλους που θα παραβιάζει την ενωσιακή νομοθεσία τις βασικές θεμελιώδεις αξίες και αρχές μας. Με πλήρη ακεραιότητα θα υπερασπιστώ τις αρχές αυτές όπως έκανα και ως αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο παρελθόν. Αυτό είναι και το εχέγγυο που κομίζω για το μέλλον. Ευχαριστώ. Συμπληρωματική ερώτηση, κύριε Σίντε. Ναι, δεν με ικανοποιεί η απάντησή σας. Γιατί το ερώτημα μου δεν αφορούσε την ενωσιακή νομοθεσία, αλλά και το κράτος δικαίου που απαιτούμε από τις χώρες προσχώρησης. Εσείς δημοσίως θα καλέσετε την Ουγγρική κυβέρνηση να ε, επιστρέψει τον Γκρούευσκι στην Βόρεια Μακεδονία ως επίτροπος. Ένα λεπτό έχετε στη διάθεσή σας κύριε Βαρχέη. Αξιότιμε ε, ευρωβουλευτά. Ε, όπως είπα, δεν πρόκειται για αρμοδιότητα δική μου. Είναι αρμοδιότητα του Επιτρόπου υπευθύνου για ζητήματα μετανάστευσης. Εγώ είμαι υπεύθυνος, θα είμαι υπεύθυνος για τις εξωτερικές δράσεις της Ένωσης. Οπότε το ερώτημα αυτό πρέπει να το απευθύνεται στον κύριο Γιώχανσον, ο οποίος θα είναι υπεύθυνο για ζητήματα μετανάστευση. Ευχαριστούμε. Για το ΕΛΚ, η κυρία Κίνγκα Γκάλ έχει το λόγο. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε υποψήφιε επίτροπε. Ε, βλέπουμε ότι είχατε μια πολύ πλούσια επαγγελματική ζωή, 25 χρόνια, ασχοληθήκατε με θέματα Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, ε, έχετε δουλέψει για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η εμπειρία σας ε, πώς θα σας είναι χρήσιμη στο χαρτοφυλάκιό σας. Ε, πώς ε, σκοπεύετε να προσφέρετε εσείς σε αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Αν έπρεπε να αναφέρω κάτι, θα έλεγα δύο πράγματα. Πρώτον, εγώ νομίζω ότι συνέβαλα στο να προσχωρήσει, να ενταχθεί η Ουγγαρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάνω εκεί ε, βάσισα και τις σπουδέ μου και την καριέρα μου. Για μένα ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία που μετά από τόσα πολλά χρόνια μπορέσαμε να επανέλθουμε στην ελεύθερη Ευρώπη. Και συνεργαστήκαμε πολύ σκληρά με πολλούς ε, συναδέλφους για να το πετύχουμε. Στην αρχή αυτό έμοιαζε πολύ μακρινή, μακρινός ε, στόχος, αλλά δέκα χρόνια χρειάστηκαν από τότε που άρχισα να δουλεύω έτσι ώστε μέχρι να μπει χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μένα αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα και είμαι περήφανος που συνέβαλα. Και έκτοτε δουλεύω ε, για μια Ευρώπη που είναι πιο ισχυρή. Και έτσι λοιπόν ε, φτάνω ε, στο δεύτερο σημαντικό μου επίτευγμα που είναι για μένα το ενιαίο δίπλωμα ευρωστεχνίας. Αυτό ήταν κάτι πολύ δύσκολο ε, προσελήφθη ναι, πολύ συγκεκριμένα γι' αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό φαινόταν ε, αδύνατο, απίθανο, αλλά τα καταφέραμε. Έμοιαζε απίθανο πολιτικά, γιατί δεν μπορούσαμε να πετύχουμε ομοφωνία από τα κράτη-μέλη, ενώ έπρεπε να υπάρχει ομοφωνία. Ήταν δύσκολο διότι υπήρχαν πάρα πολλά οικονομικά συμφέροντα, αλλά μπορέσαμε να τα ξεπεράσουμε και ήταν δύσκολο γιατί ε, είναι ένα πολύ περίπλοκο θέμα ε, τόσο από πλευράς ε, θεσμικής όσο και τεχνικής γνώσης. Είμαι λοιπόν υπερήφανος για αυτά τα δύο με τα οποία νομίζω ότι και εγώ συνέβαλα στην Ευρώπη. Η κυρία Κινγκαγκάλ, συμπληρωματική ερώτηση. Παρά κάποιες ερωτήσεις που τέθησαν, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι που το είπατε, αλλά θέλω να το, μας το ξαναπείτε. Εσείς πώς ε, αυτοπροσδιορίζεστε, ε, εντάσσεστε μέσα σε μια ομάδα, αρμονικά. Έχω και άλλη επιλογή, τι να κάνω. Αν δείτε λιγάκι τη σταδιοδρομία μου, θα διαπιστώσετε ότι ε, ανέλαβα να ε, κάνω πράγματα που δεν θα μπορούσα να τα κάνω μόνος μου. Άρα δηλαδή πάντα δούλευα μέσα σε ομάδες, είτε στην ε, Ουγγρική Διοίκηση από την αρχή της καριέρας μου, είτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε στην μόνιμη αντιπροσωπεία της χώρας μου. Ε, δεν μπορεί κανείς να δουλέψει χωρίς ισχυρή ομάδα και πάντα ήμουνα υπερήφανος για τις ομάδες ε, στις οποίες δούλεψα. Η δική μου η ομάδα αυτή τη στιγμή στη μόνιμη αντιπροσωπεία είναι κάτι για το οποίο είμαι πάρα πολύ περήφανος. Έχουμε τους σωστούς ανθρώπους που κάνουν τη σωστή δουλειά, άνθρωποι που μπορούν να δουλέψουν κάτω από πίεση, ε, που μπορούν να επιτελέσουν δύσκολα καθήκοντα, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθούμε να δουλεύουμε ενωμένοι. Και γι' αυτό, αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Δεν είμαι εγώ που ε, εκπροσωπώ την Ουγγρική Αντιπροσωπή ως πρέσβης, που δουλεύω εκεί βέβαια, αλλά εκπροσωπώ όλη την ομάδα και είμαι υπερήφανος γι' αυτό. Ευχαριστώ για την ΚΟΕ. Ο Στέλιος Κούλογλου έχει το λόγο. Εδώ είμαι, εδώ είμαι. Ας μιλήσουμε για αυτό το παιχνίδι της ανεξαρτησίας. Όπως γνωρίζουμε, προταθήκατε από την Ουγγρική κυβέρνηση, από τον κύριο Ορμπάν να λάβετε αυτή τη θέση, έτσι. Και σας ρώτησαν επανειλημμένα και άλλοι συνάδελφοι περί της υποθέσεως Γκουρεύσκη και των σχολείων της Ουγγρικής κυβερνήσεως και είπατε ότι είμαι ανεξάρτητος. Είμαι ανεξάρτητος. Εφόσον είσαστε ανεξάρτητος, γιατί δεν παίρνετε μια θέση επ' αυτών των ζητημάτων. Συγκεκριμένα, για το θέμα Γκρουεύσκη για τη Βόρεια Μακεδονία, για το άσυλο, για τα σχόλια που έκανε η Ουγγρική κυβέρνηση. Ήσασταν εξάρτητος, λοιπόν πάρτε θέση. Κύριε υποψήφιε επίτροπε, για ένα δίλεπτο. Πήρα θέση. Θεωρώ ότι η θέση μου είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επ' αυτού είναι ότι η χορήγηση ασύλου εμπίπτει στην αρμοδιότητα του κράτους μέλους. Αν δείτε, πριν αυτό πρέσβευε για την υπόθεση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα ξεκολουθώ να περασπίζουμε αυτή τη γραμμή. Η δική μου ανεξαρτησία νομίζω ότι εξυπηρετείται καλύτερα από το να ακολουθώ την ευρωπαϊκή γραμμή από αυτού. Δεύτερον, όπως εξήγησα, αυτό δεν είναι κάτι που εμπίπτει στο δικό μου χαρτοφυλάκιο. Θα ήταν δυσδυτικό για μένα πανεβατικό αν τοποθετούμεν επί των άλλων συναδέλφων. Θα αντέβαινε την αρχή της συλλογικότητας και της τρόπου επιμερισμού των καθηκόντων εντός Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συμπροματική ερώτηση, κύριε Κούλογλου. Καλώς. Σε περίπτωση που στο μέλλον, στο χαρτοφυλάκιό σας, τα καθήκοντά σας, η Ουγγαρία ακολουθεί μια στάση αντίθετη με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πάρετε θέση κατά της Ουγγρικής κυβέρνησης. Απάντηση. Δεν θα έχω επιλογή παρά να τοποθετηθώ και να υπερασπιστώ τι αξίε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω και τη γραμμή τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω εναντίον ιασδήποτε κυβερνήσεω, οδήποτε θεσμού ή ουδήποτε ατόμου. Για τους ε, σοσιαλιστές η κάτι πηρε Έχει το λόγο. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, τα τελευταία πέντε χρόνια ήσασταν ο πρέσβης της Ουγγαρίας εδώ στις Βρυξέλλες και σίγουρα σας ζητήθηκε πολλές φορές ε, η συμβουλή σας από την κυβέρνηση την οποία εκπροσωπούσατε. Για ποιο λόγο λοιπόν δείχνει η Ουγγρική κυβέρνηση τέτοια αιμονή για να πάρει το χαρτοφυλάκιο της διεύρυνσης και της γειτονίας. Καθώς ο ρόλος του Επιτρόπου αυτού απαιτεί αφοσίωση και προσήλωση στις ευρωπαϊκές αρχές και θα κληθεί να δράσει ως εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στι χώρε τη διεύρυνση. Εσεί μπορείτε να μα εξηγήσετε γιατί η Ουγγαρία επιδεικνύει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον να πάρει δικό τη υποψήφιο αυτό το χαρτοφυλάκιο. Κύριε υποψήφιο επίτροπε, είναι δύσκολο το ερώτημα, γιατί εγώ ξέρετε δεν εκπροσωπώ την Ουγγρική κυβέρνηση. Εγώ εκπροσωπώ τον εαυτό μου και μόνο εδώ ενώπιον σα. οπότε δεν μπορώ να σα απαντήσω για ποιο λόγο θεώρησε η Ουγγρική κυβέρνηση ότι είναι τόσο σημαντικό το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Αυτό που μπορώ να σα πω όμω είναι πώς και με ποιον τρόπο ένας Ούγγρος μπορεί να συμβάλλει στο χαρτοφυλάκιο αυτό και ποιες είναι οι ειδικέ γνώσεις τις οποίες μπορεί να κομίσει ένας Ούγγρος. Όπως γνωρίζετε, και εσείς ε, έχετε ουγγρική καταγωγή, ε, είμαστε γείτονε με την περιοχή της διεύρυνσης και της ανατολικής γειτονία και έχουμε στενές σχέσεις με την ε, περιοχή της γειτονία. Και η Ουγγαρία διατηρεί καλές σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής. Ίσως από αυτή τη σκοπιά μπορεί να συμβάλλει ένας Ουγγρος Επίτροπος ακολουθώντας μια παρόμοια στάση έχοντας δηλαδή και επιδιώκοντας φιλικές σχέσεις με όλες αυτές τις χώρες, κάτι που μπορεί να αποβεί προς όφελος συνολικά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Συμπληρωματική ερώτηση, κάτι Ωραία. Εντάξει. Οπότε αφού μιλήσαμε για ουγγρικές υποθέσεις και αφού μιλάμε για ουγγρικές υποθέσεις, ας συνεχίσω στα ουγγρικά. Παρακαλώ βάλτε τα ακουστικά σα. Συνάδελφοι, γιατί θα μιλήσω ουγγρικά. Εσείς θα ελέγχετε ότι εξασφαλίζεται η ελευθερία του τύπου, ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη και ότι καταπολεμάται η διαφθορά στι χώρε τη διεύρυνση τα θέματα αυτά, ποια είναι η άποψή σα για τη χώρα την οποία γνωρίζετε καλύτερα. Τι συμβαίνει ω προ αυτά τα ζητήματα στη δική σα χώρα, την Ουγγαρία. Κύριε Βαρχέη, ένα λεπτό. Δεν είναι καθήκον μου ως Επιτρόπου να αξιολογήσω τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι αρχές του κράτους δικαίου στην Ουγγαρία. Υπάρχουν δύο ε, μέλη της Επιτροπής, ο κύριος Ράιντας και η κυρία Γιούροβα, ε, που θα είναι αρμόδια για τα ζητήματα αυτά και νομίζω ότι με συναδελφικότητα και με ε, ορθή στάση από την πλευρά μου θα πρέπει εκείνοι να τεθούν επικεφαλής μιας τέτοιας αξιολόγησης και είμαι βέβαιος ότι θα το πράξουν οι δύο επίτροποι αυτοί. Next green εκ μέρους των πρασίνων, παρακαλώ, όλοι μας ε, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ε, όσον αφορά το κράτος δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι αξιόπιστη και να μην αμφισβητούνται οι αποφάσεις της. Ε, ε, στις γραπτές σας απαντήσεις λέτε ότι δεν πρέπει να γίνει επιλογή ανάμεσα στα εθνικά και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Όμως η διαδικασία του άρθρου 7 κατά τη Ουγγαρίας μας έδειξε ότι μερικές φορές δεν, είναι, δεν συμφιλαιώνονται αυτοί, αυτοί οι δύο στόχοι. Όταν αναφερθήκα στην ε, ε, Ουγγαρία, ε, σχεδόν απορρίψατε όλες τις κατηγορίες κατά της Ουγγαρίας και σχεδόν είπατε ότι η νίκη του Όρμπαν δεν δημιουργεί πρόβλημα στο κράτος δικαίου στην Ουγγαρία. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ το ψήφισμα και το όλο σκεπτικό πίσω από το ψηφίσμα, κατ' ουσίαν εκφράζουν τις δικές σας τις απόψεις για να κρίνετε υποψήφιες χώρες σχετικά με το αν τηρούν το κράτος δικαίου ή όχι. Και αν όχι, τι μπορείτε να μας πείτε, μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι τα κριτήρια της Κοπενχάγης δεν θα αντικατασταθούν από τα κριτήρια της Βουδαπέστης. Ε, στην εισαγωγή μου, ε, στην ομιλία μου είπα ότι είναι απαραίτητο να έχουμε σύνθεση των εθνικών συμφερόντων ε, να τα συνδυάζουμε αυτά με τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Και αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αλληλοεξαιρούνται. Η δική μου η προσέγγιση είναι ότι τα ευρωπαϊκά συμφέροντα βασίζονται πάντα στα συμφέροντα των κρατών μελών. Ε, Βεβαίω η τέχνη εδώ είναι να αναζητηθεί ένας κοινό δρόμος αποδεκτός για όλους. Στους τομείς ε, που θα κληθώ να εργαστώ εγώ δεν μπορώ να εργαστώ χωρίς να υπάρχει σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις η ομόφωνη υποστήριξη από τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να εργάζομαι έχοντας αυτό κατά νου, αλλά είμαι συνηθισμένος να το πράττω, γιατί το χαρτοφυλάκιο που σας ανέφερα, που δούλευα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαιτούσε κάτι τέτοιο. Δεν φοβάμαι όμως να κάνω επιλογές και αυτές οι επιλογές σαφώς και βασίζονται στα κριτήρια της Κοπενχάγης, τα οποία δεν μπορούν να νοθευτούν ε, να διευρυνθούν από ένα και μόνο επίτροπο. Εγώ δεν την έχω αυτή τη δύναμη και δεν θέλω καν να την έχω. Τα κριτήρια της Κοπενχάγης εξακολουθούν να αποτελούν τη βάση οποιασδήποτε διαδικασίας διεύρυνσης και εγώ θα μεριμνήσω έτσι ώστε να γίνονται απολύτως σεβαστά σε όλες τις χώρες που ενδιαφέρονται για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμπληρωματική ερώτηση παρακαλώ έχοντας κατά νου ε, την αφοσίωσή σας στην Ουγγρική κυβέρνηση μέχρι τώρα, επιτρέψτε μου να επιδιώξω μια πιο πιστική απάντηση από πλευρά σας. Για να δούμε. Πιστεύετε ότι ένα κράτος το οποίο ε, καταπιέζει την αντιπολίτευση, σχεδόν ελέγχει πλήρως ε, τα μέσα ενημέρωσης, ε, ε, εξωθεί ανθρώπους ε, στην σύνταξη, είναι διακριτικό έναντι μειονοτήτων. Πιστεύετε ένα κράτος πληρεί τα κριτήρια για ένα κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν οποιαδήποτε χώρα που επιθυμεί την ένταξη βρισκόταν με τέτοιου είδους ελλείψεις, προφανώς ε, δεν θα μπορούσα να επιτύχω την υποστήριξη των κρατών μελών για να ε, δεχτούν μια τέτοια χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου η δική μου δουλειά θα βασίζεται στη δουλειά του προκατόχου, δηλαδή ε, να διεκδικούμε ένα σωστό ε, σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με ανεξάρτητη δικαιοσύνη, με καταπολέμηση της διαφθοράς, με ανεξάρτητους δημοκρατικούς θεσμούς, όπου θα γίνονται έλεγχοι, θα επιδιώκονται ισορροπίες, οτιδήποτε δηλαδή απαιτείται ε, στο πλαίσιο μιας διεύρυνσης. Να είστε λοιπόν σίγουροι ότι ε, αυτές τις αρχές θα υπηρετήσω και όσον αφορά τις ενταξιακές χώρες. Ευχαριστώ κύριε Βερχέη. Πάμε στην ομάδα Renew Europe. Κυρία Φονβίζα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Υποψήφια Επίτροπε, και ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα. Η εκλεγή σαν πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η κυρία Βαντερ Λάιν, δήλωσε στην αποστολή που σα ανέθεσε ότι συνεργάζεται στενά με τον ύπατο εκπρόσωπο για τι σχέσει με την Τουρκία. Αναφερθήκατε εν παρόδο στην Τουρκία, αλλά οι ενταξιακέ επεμβατεύσει τη Τουρκία έχουν ουσιαστικά αποτελματωθεί και άλλα κεφάλαια ε, δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι ανοίγουν ή κλείνουν, ενώ η Τουρκία εξακολουθεί να απομακρύνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα όρο για ένταξη μια υποψήφια χώρα είναι ο σεβασμό ε, κοινών αξιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και δέσμευση να τη προωθεί. Όπω ακούσαμε, αυτά τα κριτήρια συμπεριλαμβάνουν τη σταθερότητα των θεσμών, εγγύηση για τη δημοκρατία, το κράτο δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα και σεβασμό και προστασία των μειονοτήτων πιο συγκεκριμένα σχετικά με αυτά τα κριτήρια. Τι βήματα θέλετε να δείτε η Τουρκία να κάνει πριν οι διαπραγματεύσεις οι ενταξιακές να μπορέσουν να ξαναρχίσουν. Ευχαριστώ. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, Τουρκία. Πρέπει να έχουμε έναν πλήρη διάλογο με την Τουρκία. Σε αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε να επιμείνουμε ε, των ενσυχιών μας είτε αφορά την ελευθεροτυπία, είτε την εξαρτησία του δικαστικού κλάδου, τη φυλάκιση δημοσιογράφων ή την οπισθοχώρηση όσον αφορά το κράτος δικαίου. Αυτά τα θέματα πρέπει να συζητηθούν και να αντιμετωπιστούν όχι μόνο στο πλαίσιο το ενταξιακό, αλλά και σε ευρύτερο πλαίσιο, διότι βεβαίω έχουν αντίκτυπο επί των σχέσεών μα με την Τουρκία. Αλλά δεν πρέπει να λησμονεί κανεί τα συμφέροντα που είναι πέραν αυτών, τα συμφέροντά μας. Φερρυπίν, Τελωνιακή Ένωση, αλλά και η σχέση μας όσον αφορά τη συνεργασία για τα μεταναστευτικά. Χρειάζεται ισορροπημένη προσέγγιση και άποψη, χωρίς να θυσιάζει καμία από τις θεμελιώδεις αξίες και αρχές που πρέπει να υπερασπιστούμε και να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε στην Τουρκία. Είναι σημαντικός ο διάλογος σχέση με την Τουρκία. Αν διαλόγου θα έχουμε όλο και μικρότερη επιρροή έναντι της Τουρκίας. Φερρυπίν. Επιρροή είναι πολύ σημαντική όσον αφορά τη χρηματοδότηση την πρωταξιακή. Δεν είχα ερώτηση επ' αυτού, αλλά παρόλα αυτά θα ήθελα να εκφράσω τη σχετική μου άποψη, διότι γνωρίζω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα για το Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο έχει συγκεκριμένη σταθερή θέση όσον αφορά την ακύρωση την υποστήριξη της πρωταξιακή στην Τουρκία. Εγώ θα ήμουν πιο προσεκτικός στην προσέγγιση μου. Ήδη έχει περικοπεί από 600 εκατομμύρια στα 250 εκατομμύρια και θέλουμε να κάνουμε περαιτέρω περικοπές και να πάμε περίπου στα 130 εκατομμύρια. Όμως αυτό είναι και ο πυρήνας της χρηματοδότησής μας και αυτή είναι μια χρηματοδότηση της κοινωνίας των πολιτών. Εάν περικόψουμε αυτή τη χρηματοδότηση θα εξαφανιστεί η κοινωνία των πολιτών από την τουρκική κοινωνία. Θα πρέπει να συνεχίσουμε ε, σε αυτό το τομέα. Κύριε Φομβίζε, συμπληρωματική ερώτηση. Ευχαριστώ. Μπορείτε να μας δώσετε κάποια σαφή παραδείγματα της δικής σας εμπειρίας όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις μεταξιακές χώρες προς ένταξη όσον αφορά τις αξίες κυρίως το κάτω δικαίου, ανθρώπινα δικαιώματα και σεβασμό και προστασία των μειονοτήτων. Κύριε Βερχέη, για ένα λεπτό. Δύσκολη ερώτηση, διότι εγώ δεν έχω πραγματοποιήσει συνταξιακέ διαπραγματεύσεις με καμία από αυτές τις χώρες, εκπροσωπούσα ένα από τα κράτη-μέλη. Βέβαια, σε αυτές τις ε, συζητήσεις, όταν προσπαθούσαμε να ε, προσμετρήσουμε τις επιδόσεις των διαφόρων προσένταξη χωρών, Αυτά τα θεμελιώδη έπρεπε να αξιολογηθούν πρώτα. Και βέβαια στην γειτονιά μας μπορούμε να αισθανόμαστε ασφαλείς μόνο αν γίνονται σεβαστές αυτές οι θεμελιώδεις αξίες και μόνιμα να γίνονται σεβαστές αυτές οι αξίες και να στηρίζονται από τους θεσμούς. Να μην υπάρχουν μόνο στα πλαίσια του νόμου με μια ευρία έννοια, Έκκλησή μου θα ήταν προς αυτές τις χώρες η εξής. Όχι μόνο να θεσπίσουν νομοθεσία κατάλληλη, αλλά αυτές οι αρχές να μπορούν να εφαρμόζονται και να λειτουργούν για το λαό τους. Ευχαριστούμε κύριε υποψήφια επίτροπε. Τελευταίο ερώτημα εκ μέρους του ΕΛΚ, ο κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ κύριε Υποψήφιο Επίτροπε. Είχα ένα ερώτημα για την Τουρκία, το οποίο μόλις σας τέθηκε και απαντήθηκε από εσάς. Οπότε, όσον αφορά την προενταξιακή διαδικασία, υιοθετείτε ε, τη θέση του ΕΛΚ ότι τα χρήματα θα πρέπει να κατευθύνονται προς την κοινωνία των πολιτών και την τουρκική συμμετοχή σε προγράμματα όπως το Erasmus+. Plus. Αυτή νομίζω ότι είναι μια συμφωνημένη γραμμή που έχουμε και σας ευχαριστούμε για αυτή την κοινή θέση ε, που έχετε με το ΕΛΚ. Να περάσω λοιπόν στα Δυτικά Βαλκάνια. Για να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίε που εξέφρασαν κάποια κράτη-μέλη όσον αφορά την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Εσείς θα εφαρμόσετε τα κριτήρια τη Κοπενχάγης με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε χώρα να κρίνεται πράγματι με βάση τις επιδόσεις τη. Μήπω η μεθοδολογία λοιπόν δεν θα πρέπει να είναι μια συμφωνία πακέτο, αλλά να εκτιμάται και να αξιολογείται η κάθε χώρα ανάλογα με τις περιστάσεις που επικρατούν σε αυτήν, καθώς και σχετικά πρόσφατες ε, υπαναχωρήσεις. Για να υπάρξει ομοφωνία στο Συμβούλιο, μήπως θα μπορούσε μόνο μία χώρα να λάβει το πράσινο φως για την ε, έναρξη των ενταξιακών της διαπραγματεύσεων, για να διατηρηθεί και αυτή η δυναμική τουλάχιστον. Κύριε Βαρέη, είναι δύσκολο και στρατηγικό ταυτόχρονο το ερώτημα που θέτεται. Η απάντησή μου είναι διτή. Πρώτον, καμία ενταξιακή ε, διαδικασία δεν μπορεί να είναι αξιόπιστη αν δεν βασίζεται σε συγκεκριμένες επιδόσεις και την αξιολόγηση αυτών. Δεν αν δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο επίτευγμα, δεν μπορεί βεβαίως και να υπάρχει ε, όφελος για την χώρα. Βεβαίως μπορεί να, σταθούμε, να βρεθούμε κάποια στιγμή σε ένα κρίσιμο σημείο όπου μία, δύο ή τρει υποψήφιε χώρες έχουν επιτύχει την εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων. Εγώ δεν έχω εκ των, υστέρων, ε, προτέρων μάλλον στάση. Αν πρόκειται για μία χώρα που τα έχει εκπληρώσει όλα, τότε είναι μία. Αν είναι δύο, δύο. Αν είναι τρεις, τότε είναι τρεις. Αλλά δεν πρέπει να εμποδίσουμε τον, καμία χώρα να επιτύχει τους στόχους που τους έχουμε θέσει. Και το μεγαλύτερο κίνητρο που μπορούμε να δώσουμε σε αυτή την κατεύθυνση είναι όσο μεγαλύτερη προθυμία δείχνουν οι υποένταξη χώρε, τόσο μεγαλύτερη προθυμία και βοήθεια θα τους, ε, θα τους παρέχουμε εμείς. Είναι λοιπόν ε, δύσκολος στόχος να, ε, να ξεφύγουμε από αυτήν την ομαδοποίηση των χωρών, όμως δεν είναι και ανέφικτος στόχος. Το, η δεύτερη πτυχή της απάντησής μου, της μου αφορά την ε, γεωπολιτική διάσταση των Δυτικών Βαλκανίων. Τα επόμενα πέντε χρόνια δουλειά μας θα είναι να δημιουργήσουμε μακροπρόθεση, μακροπρόθεσμη, μακρόπνοη ευμερία, σταθερότητα και δημοκρατία. Βεβαίως, το να επιλέξουμε μία ή μόνο δύο χώρες ε, για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων θα έχει αντίκτυπο. Αυτό ε, θα πρέπει να το έχουμε ως ε, στοιχείο υπόψη μας όταν λαμβάνουμε, θα λάβουμε τις σχετικές αποφάσεις. Κύριε Γκάλερ, συμπληρωματική ερώτηση. Ναι, βεβαίω, προφήτε δεν είμαστε. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε για το πού θα, θα, θα βρισκόμαστε σε πέντε χρόνια. Αν όμω εναπόκειτο σε εσά να αποφασίσετε. Πώς θεωρείτε, πόσο χρόνο θεωρείτε ε, ότι θα χρειαστεί για τη διαπραγμάτευση. Για την Κροατία ήταν 8 χρόνια, για παράδειγμα. Ε, τα επόμενα 5 χρόνια μπορεί να ενταθούν οι διαπραγματεύσει χωρί όμω να καταλήξουν σε προσχώρηση, προσχώρηση κάποια χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε λοιπόν τις φιλόδοξες αυτές χώρες ε, να τους παράσχουμε κίνητρα με στοιχεία, με μέσα που θα υπερβαίνουν τις εμπορίες, ε, της ε, Συμφωνίας Εμπορικών ε, Συναλλαγών. Υποψήφιος Επίτροπος, σε πέντε χρόνια σκοπός μου είναι να έχουμε πιο ανεπτυγμένα Δυτικά Βαλκάνια, να έχει επιτευχθεί ειρήνη μεταξύ Κωσυφοπεδίου και Σερβίας, να έχει απαλλαγή πλήρως το Κόσοβο από τις θεωρήσεις και να έχουν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Αλβανία και την Βόρεια Μακεδονία και ενδεχομένως να έχουν ολοκληρωθεί, μάλιστα να βρίσκονται στο τελικό τους στάδιο και να ε, βρεθεί σε αντίστοιχα προηγμένο στάδιο και η Σερβία. Αυτός, αυτό είναι το όραμά μου για το που θέλω να, να βρεθούμε σε πέντε χρόνια. Ε, μπορεί να ακούγεται πολύ φιλόδοξο, αλλά χωρίς φιλοδοξία, ξέρετε, πολλές φορές δεν επιτεχάνονται και οι στόχοι. Όσον αφορά την ανατολική εταιρική σχέση, η προσέγγιση μου για τις, χώρες, ε, ε, για τις τρεις εκείνες χώρες με τις οποίες έχουμε υπογράψει ε, συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, το μήνυμά μου είναι αν θέλουμε να κάνουμε περισσότερα, θέλουμε και εμείς να κάνουμε περισσότερα. Και μπορούμε να εντάξουμε και στην καθημερινότητά μας αυτή την πρακτική και αυτή τη διαδικασία. μέσα τη πράσινη συμφωνία, μέσω τη ψηφιακή οικονομία, μέσω των μεταφορών και τη ενέργεια υπάρχουν μια σειρά από τομεί στου οποίου μπορούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία μα. Ευχαριστώ σα συνάδελφοι για τι ερωτήσει. Ευχαριστώ και τον υποψήφιο επίτροπο που απάντησε σε όλε τι ερωτήσει. Κύριε Βερχέη, να δώσω ξανά το λόγο σε εσά για μια σύντομη ομιλία σας για περίπου 5 λεπτά. Πρόεδρε, εξότιμα μέλη, ευχαριστώ όλους σας για ανοιχτή και ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων. Σαφέστατα θέσατε επιτάπητο στις προτεραιότητές σας σχετικά με τη διεύρυνση και την πολιτική γειτονία και το σχετικό χαρτοφυλάκιο. Διευκρινίσατε επίσης τις προσδοκίες σας από μένα αν αποφασίσετε να εγκρίνετε το διορισμό μου. Ε, ακούσαμε ήδη τις προτεραιότητες μου και ελπίζω τώρα στο τέλος των συζητήσεών μας ότι μοιραζόμαστε την άποψη ότι υπάρχει ε, μια γενική σύγκληση στους στόχους μας θα πρέπει να ενισχύσουμε την διαδικασία διεύνησης και να ενισχύσουμε μια αξιόπιστη ευρωπαϊκή προπτική για τα Δυτικά Βαλκάνια. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε αυτά αποτελέσματα βραχυπρόθεσμα για τους λαούς των, της γειτονιάς μας, για την καθημερινή τη ζωή τους μέσω οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό θα αυξήσει το ρόλο μας και την επιρροή μας θα πρέπει να έχουμε επαρκείς οικονομικούς πόρους στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο για να υποστηρίξουμε τους στόχους μας τη πολιτικής μας. Όλες οι προσπάθειες θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν πλήρω και να εξυπηρετούν τις αξίες μας και τα συμφέροντά μας είτε στα Δυτικά Βαλκάνια, στους, Ανατολικού στους ανατολικούς εταίρους ή στην νότια γειτονιά μας. Πιστεύω ότι αυτή είναι μια εξαιρετική βάση συνεργασίας. Είμαι αποφασισμένο να συνεργαστώ στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με τα μέλη αυτή τη επιτροπή ιδιαίτερα. Έτσι δε περαιτέρω βλέπω σημαντική συμπραγματικότητα μεταξύ των ρόλων μα. Η κοινοβουλευτική διπλωματία και οι σχέσει με τι ε, κυβερνήσει. εγώ θα βασίζομαι να τα χρησιμοποιήσω αυτά πλήρω προ συμφέρον τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Θα παράσχω κάθε αναγκαία υποστήριξη προς εσάς για να εργαστείτε αποτελεσματικά. Τέλος. για την επέτειο ενός γεγονότος θέλω να μιλήσω τώρα που διαμόρφωσε η σημερινή Ευρώπη. Πριν από 30 χρόνια, 9 Νοεμβρίου 1989, έπεσε το τείχος του Βερολίνου. Άνοιξε έτσι ο δρόμος για την επανένωση της Γερμανίας και την επανένωση της Ευρώπης. Ιστορική ευκαιρία και η Ευρώπη και οι ηγέτες Ευρώπης ήταν πολύ γενναίοι να εκμεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία. Δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν προφανές. Πολλοί είχαν αμφιβολίες. Τι γίνεται με τους κινδύνους. Προσπαθήσανε να επιβραδύνουν τα γεγονότα, αλλά η ιστορία απέδειξε ότι έσφαλαν. Σήμερα είμαστε όλοι ευγνώμονες προς εκείνους που κατέστησαν αυτό εφικτό. Σήμερα γνωρίζουμε ότι ήταν προς γενικό ευρωπαϊκό συμφέρον να καταρρεύσει ο τείχος και να διαδοθεί η δημοκρατία, ευημερία και το κράτος δικαίου μέσω Ενωμένης Γερμανίας και Ενωμένης Ευρώπης. Είναι μια τεράστια επιτυχία, όμως δεν είμαστε ακόμα στο τέλος του δρόμου. Πρέπει να συνεχίσουμε τη διάδοση της ευημερίας, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στο κέντρο της Υπήρου μας και στα Δυτικά Βαλκάνια είναι προς συμφέρον τους, είναι προς συμφέρον μας. Έχουμε μια ιστορική ευκαιρία επ' αυτής της θητείας να εφαρμόσουμε μια μακροκρόνια ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία σε μια περιοχή που δεν τα έχει δει αυτά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν θα χάσουμε αυτή την ιστορική ευκαιρία. Ούτω ώστε 30 χρόνια από σήμερα μπορούμε να κοιτάξουμε υπερηφάνεια προς το παρελθόν και να πούμε Είμαστε άξιοι των προκατόχων που οικοδόμησαν την Ευρώπη και εμείς παίξαμε τον ρόλο μα. Δεν θα διστάσουμε πλέον να βοηθήσουμε τους γειτονέ μας να του πλησιάσουν, να τους στείλουμε το χέρι βάσει των, της αξίας τους και των επιθυμιών τους. Θα εργαστώ επ' αυτού και θα ήθελα να είμαι εταίρος σας ούτως ώστε αυτό να συμβεί. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Κυρίε και κύριοι, ευχαριστούμε του φιλοξενούμενους μα που συμμετείχαν σημερινή συνεδρία. Ευχαριστώ του συναδέλφου που έθεσαν πολύ ενδιαφέρουσε ερωτήσει και όλου του συναδέλφους που τήρησαν το χρόνο που του διετέθη. Αυτό μα βοήθησε πάρα πολύ. Και τέλο να ευχαριστήσω εκ νέου, εκ μέρου τη Επιτροπή μα, τον κύριο Όλιβε Βαϊχέη που ήταν εδώ μαζί μα, περίπου τρει ώρε απαντούσε στι ερωτήσει μα, πέρα στη συνεδριά σα. Σα ευχαριστώ πολύ. Γεια σα.